μόνο σύνολο δικαιωμάτων υπέρ των καταναλωτών. Δεύτερον, σε ε, Μικρο, σε, επίπεδο, σε, μικρό επίπεδο πρέπει να αποσυμμακρύνουμε αυτά τα, αυτούς τους φραγμούς που έχουν τοποθεθεί εσκεμένα ανάμεσα στους επιμέρους καταναλωτές και στην άσκηση της, ε, ε, του δικαιώματος της επιλογής γνωρίζοντας όμως όλα τα στοιχεία και όντα ενημερωμένοι. Τα εμπόδια ε, στη νομική νομική βεβαιότητα, στην ε, ε, πολύπλοκη τιμολόγηση και μένα πολύπλοκη τιμολόγηση, ε, στην αλλαγή των όρων των συμβάσεων κτλ. Ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύσουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία λείπουν στον χώρο τη αγορά, όπω για παράδειγμα το καλύτερο επίπεδο προστασία των καταναλωτών και το δικαίωμα για συλλογική αποζημίωση. και για του επιχειρηματίε και για του καταναλωτέ, θέλουμε μέσα από την εργό συμμετοχή να δώσουμε και στους δύο όλα τα ωφέλη τη εσωτερική αγορά. Θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια αν η αγορά είναι φιλική προ το χρήστη. Κατά την άποψή μου, οι, οι, οι μεταρρυθμίσεις τη τη αγοράς της θα πρέπει να οδηγήσουν στην οικοδόμηση μια αγορά ε, που να είναι φιλική προ το χρήστη. Ανεξάρτητα ποιοι είναι, ποιοι είναι οι χρήστε. Καταναλωτέ, μικρομεσαίες επιχειρήσει, επιχειρήσει ε, offline ή, ε, και online. Αυτό σημαίνει ένα και μόνο σύνολο κανόνων. Πρόσβαση στα δικαιώματα στο σημείο πώληση. Διαφανή παρακολούθηση τη αγορά. Αξιόπιστη ανάλυση τη αγορά. Ε, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων. Μελέτες, ε, στοχοθετημένες μελέτες αποτυχίας της αγοράς και, ε, και καταναλογία σωστές αποζημιώσεις για να επαναξεκινήσουμε την εσωτερική αγορά στην ψηφιακή, ε, στην ψηφιακή εποχή, χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο δικαιωμάτων, δασμών, ε, εφαρμογής και προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να αλλάξουμε από την οτροπία της ρύθμισης και να εστιάσουμε τις, τις προσπάθειές μας στα αποτελέσματα της αγοράς. Στόχος καλύτερες τιμές και, και καλύτερη επιλογή και για τους καταναλωτές αλλά και για τα νοικοκυριά με ένα σύγχρονο ενιαίο σύνολο κανόνων που να βασίζεται σε ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο προστασίας. Από τότε που παρουσιάσαμε την πρότασή μας, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, υπήρξε σημαντική βαθμό ε, βαθμός συζήτησης για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, μεγάλος προβληματισμός. Άκουσα όλε τι πλευρέ. Παρατήρησα ότι υπάρχει υποστήριξη για την πρόταση, αλλά ταυτόχρονα έγιναν και πολλά κριτικά σχόλια από αυτού που φοβούνται ότι η πρόταση θα μειώσει το επίπεδο προστασία των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σα πω ότι αντιμετωπίζω αυτέ τι επικρίσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ειλικρινά ότι η μελλοντική οδηγία θα πρέπει και πράγματι θα πράξει θα ωφελήσει όλα τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο το απόγευμα η Επιτροπή σας έχει διοργανώσει μία ακρόαση για την πρόταση οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν έχω καμία αμφιβολία για τα αποτελέσματα αυτή τη ε, ακρόαση που θα είναι ιδιαίτερα καρποφόρα. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε τι απόψει ε, του νέου εισηγητή, του Αντρέα Σουάμπ, τον οποίο θα ήθελα να τον συγχαρώ, γιατί ανέλαβε αυτό το τόσο σημαντικό καθήκον. Αλλά επιτρέψτε μου να εκφράσω ορισμένε σκέψει μου εδώ. Πρώτα απ' όλα, Ακούγοντας τις επικρίσεις ε, ε, της πρότασης, ε, φτάνω στο συμπέρασμα για το ότι πολλοί εξακολουθούν να αισθάνονται αβεβαιότητα όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά ήδη η αξιολόγηση αντικτύπου που ενέχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει πολλέ από τι ανησυχίε αυτέ. Προβλέπει μια ανάλυση σε βάθο ε, όσον αφορά τι ανεπάρκειε ε, τη πρότασή μα και δεσμεύομαι να συνεχίσουμε την εργασία περαιτέρω. Ιδιαίτερα στο άμεσο μέλλον θα ε, υποβάλω μια επιπρόσθετη ποιοτική μελέτη όσον αφορά το πόσο ο καταναλωτής βλέπει τις διαθέσιμες ε, δυνατότητες αποζημίωσης για τα, ε, για τα ελαττωματικά αγαθά. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη. Δεύτερον, έχουν αναφερθεί διάφορες ανησυχίε όσον αφορά το εύρο της πρότασης. Οι υπηρεσίε μου έχουν προετοιμάσει ένα συγκριτικό πίνακα, ο οποίο δείχνει τον αντίκτυπο των βασικών στοιχείων τη πρόταση στα Τη πρόταση στα εθνικά επίπεδα τη ε, προστασία του καταναλωτή. Επίσης, διατυπώθηκε και, ένα συνοδευτικό σημείωμα, το οποίο ασχολείται με τα βασικά ε, νομικά ζητήματα, τα οποία κρεμούν και τα οποία έχουν ε, αναφερθεί μέχρι στιγμής. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συγκριτικό πίνακας δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει την αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά είναι, ε, είναι συμπληρωματικός της αξιολόγησης αντικτύπου είναι ένα έγγραφο ενδεικτικό το οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω, ε, περαιτέρω επεξεργασία. Η παρούσα έκδοση του πίνακα δείχνει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, η πρόταση μειώνει την προστασία του καταναλωτή. Αντίθετα, έχουμε περισσότερα δικαιώματα όσον αφορά ε, την, την, την παράδοση, τα, ε, ε, κρυμμένα, ε, τις κρυμμένες χρεώσεις, την περίοδο, μεταβατική περίοδο 14, 14 ημερών και για πρώτη φορά απαγορεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα, απαγορεύονται τα έντυπα με με προσυμπληρωμένα σημεία. Επίσης προστασία όλων των συμβάσεων εκτός των εγκαταστάσεων πώλησης. Λαμβάνοντα υπόψη και τι απόψει των ε, οργανώσεων των καταναλωτών, των εθνικών αρχών αλλά και των άλλων εμπλεκομένων, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κατανοητέ και θεμητέ ανησυχίε για το σωστό επίπεδο προστασία, για παράδειγμα σε σχέση με την περίοδο εγγύηση ή ε, με τι αποζημιώσει. Είμαι έτοιμη να, εργαστούμε, να συνεργαστούμε περαιτέρω προ την κατεύθυνση αυτή και μαζί σα και με το Συμβούλιο για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να δούμε ποια δικαιώματα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Όμως πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι έτοιμη να ε, υποχωρήσω σε σχέση με αυτό που είπαμε. Ενιαίο σύνολο ε, ε, κανόνων που να ισχύει για όλους. Από το μικρό κατάστημα μέχρι την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή είμαι σίγουρη ότι μέσα από τις διαπραγματεύσεις θα μπορέσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία με σκοπό το συμφέρον των καταναλωτών, των Ευρωπαίων καταναλωτών για τα επόμενα χρόνια. Σας διαβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή ε, στις επικοδομητικές συνεισφορές. Επίση, χάρη σε ένα νέο σύνολο ενιαίων ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, θα μπορέσουμε να εργαστούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι ε, γνώσει των καταναλωτών για τα δικαιώματά του στο σημείο πώληση τα, δικαιώματα των καταναλωτών δεν είναι άχρηστα αν δεν τα γνωρίζουν οι ίδιοι οι καταναλωτές. Ε, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτέ αλλά και πολύ συχνά και οι έμποροι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Και εδώ ε, θέλουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι υπηρεσίε μου έχουν αρχίσει την προετοιμασία νέων πρωτοβουλειών και ε, θα καλέσουμε όλες τις όλους τους εμπειρογνώμονες ε, επιτόπου για να προσδιορίσουμε όλοι μαζί τις ε, βέλτιστες πρακτικές λύσεις που να είναι και, απο, αποτελεσματικές από άψη κόστους ωφέλους. Και τώρα φτάνω στο επόμενο θέμα. Τα ουσιαστικά δικαιώματα είναι σημαντικά μόνο όταν συνοδεύονται από σωστή εφαρμογή και από αποτελεσματικές αποζημιώσεις των καταναλωτών. Και τώρα επιτρέψτε μου να ασχοληθώ με τα δύο αυτά ζητήματα. Παρατηρούμε ότι Όσο επεκτείνονται οι αγορές, ε, πλήττονται οι ομάδες των καταναλωτών από ε, τις ίδιες παράνομες πρακτικές των εμπόρων, ε, παραπλανητική διαφήμιση, διανομή και πώληση προϊόντων που δεν είναι ασφαλή, υπερχρέωση των πελατών, παράληψη κρίσιμης πληροφορίας είναι σίγουρο ότι με βάση του υφιστάμενου κανόνε και τι πρακτικέ ε, στα κράτη-μέλη, πολύ συχνά οι καταναλωτέ δεν, δεν παίρνουν τη σωστή αποζημίωση. Εξετάζουμε το θέμα αυτό σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αναθέσαμε μελέτε, συζητήσαμε το ζήτημα με όλου του εμπλεκόμενου, κάναμε έρευνε, δημόσιε διαβουλεύσει και οι υπηρεσίε μου τώρα εργάζονται προ την κατεύθυνση τη αξιολόγηση αντικτύπου με σκοπό την ε, αξιολόγηση των πιθανών λύσεων. Το είπα και προηγουμένω και θα ήθελα να το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νοοτροπία έγερσης αξιώσεων στην Ευρώπη. Οι μηχανισμοί με τις σωστές δικλείδες ασφαλείας κατά της κατάχρησης και που να συνεπάγονται ελάχιστο κόστος για όλους τους εμπλεκόμενους, αυτά είναι τα βασικά μας μελήματα. Και τέλος θα ήθελα ε, να σας εκφράσω ορισμένες σκέψεις μας για την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως είπε και ο Μάλκο. Ο πρόεδρος Μπαρόζο πρόσφατα είπε ε, ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δώσει πολλά δικαιώματα στους πολίτες της, ε, εξακολουθεί να παραμένει πρόκληση η εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών. Τι σημαίνει ότι οι πολίτες θα πάρουν στην πράξη τα δικαιώματα που έχουν θεωρητικά. Και εδώ πρέπει να, και από τότε που ανέλαβα τα, ε, τα καθήκοντά μου, εργάστηκα ιδιαίτερα προ την κατεύθυνση αυτή. Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια ε, νέα διάσταση συντονισμένη ε, πανευρωπαϊκή εφαρμογή με τα λεγόμενα SWIPs, τα οποία έχουμε ε, εφαρμόσει σε στενή συνεργασία με τι Εθνικέ Αρχέ το 2007. Παρόμοια, κατά τον ίδιο τρόπο, εξετάσαμε προσεκτικά ιδιαίτερου κλάδου τη αγορά, αεροπορικέ μεταφορέ, κινητή τηλεφωνία και ηλεκτρονικά αγαθά, για να δούμε κατά πόσο υπάρχει με του κανόνε υπέρ των καταναλωτών. Και όπου εντοπίστηκαν προβλήματα και δεν διορθώθηκαν γρήγορα, τότε ε, ξεκινήσαμε δράση κατά των ε, παραβατών. Το αποτέλεσμα αυτών των sweep, των sweeps είναι μια καινοτομία, καινοτόμο μέθοδος εφαρμογής. Διότι με τον τρόπο αυτό αποστέλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους εμπόρους, δηλαδή ότι ε, όλα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα μέτρα ε, κατά ενός κράτους μέλους, αλλά αντίθετα δεν υπάρχει ε, ένας παράδεισος, ασφαλής παράδεισος που να τους βοηθά να ε, αποφύγουν την αποτελεσματική εφαρμογή. Τώρα, όσον αφορά την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή του Ιουλίου, καθορίζονται βασικοί κανόνε προτεραιότητα που θα δώσουν το συνολικό πλαίσιο για την ε, πολιτική εφαρμογή των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια. Οι προτεραιότητε αυτέ ε, συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων καλύτερη παρακολούθηση τη αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εντοπίζονται οι αγορέ που δεν ανταποκρίνονται τι προσδοκίε των καταναλωτών, η ανάλυση των τάσεων, επίση η ισχυρότερη συνεργασία για την εφαρμογή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, με τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα Κίνα και Ηνωμένε Πολιτείε, καλύτερη ε, περισσότερη διαφάνεια ε, και ορατότητα όσον αφορά τους ελέγχους και τώρα όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένη δράση. Η άποψη και η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό είναι κρίσιμη σημασία για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής προς την κατεύθυνση εφαρμογής των νόμων στα επόμενα χρόνια. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας, εδώ τελειώνει η παρέμβασή μου και ελπίζω να μας υποστηρίξετε στις πρωτοβουλίες μας και με τη σειρά μου σας διαβεβαιώνω ότι θα λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη όλες τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you uh, very much indeed, Commissioner. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ήταν, ήσασταν χαρακτηριστικά σαφείς και μας παρουσιάσατε όλο το πρόγραμμά σας ε, για τα ζητήματα που άπτονται των καταναλωτών με εξαιρετική σαφήνεια. Ε, νομίζω ότι θα σας έχουμε ακόμη περίπου 40 λεπτά μαζί μας, αν δεν κάνω λάθος. Να σας πω ποιοι είναι οι ομιλητές. Ε, θα πρέπει να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας, γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος. Uh, and Mrs. Mrs. Mr. Mr. Rochefort, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο να εγγραφεί στον κατάλογο. Όλοι θέλουν να σα μιλήσουν, Επίτροπε. Ε, παρακαλώ να είστε σύντομοι και θα ακούμε τι παρεμβάσει ανά γιατί γίνεται καλύτερο διάλογο έτσι. Άντριος Φαμπο, μα για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ε, καθώ ζήτησαν πολλοί συνάδελφοι το λόγο, θα είμαι σύντομο. Καταρχήν, ε, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κούνεβα, για την παρουσίασή σας. και έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι ε, κατά τη θέσπιση της νομοθεσία στην Ευρώπη για την προστασία του καταναλωτή βρισκόμαστε πράγματι εδώ, όπως είπατε και εσείς σε ένα turning point, σε ένα σημείο καμπή. Όμω, ε, θα πρέπει σε αυτό το σημείο καμπή πράγματι να θέσουμε και τι σωστέ προτεραιότητε, τα πράγματα δηλαδή όπως πρέπει σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών και γι' αυτό θα πρέπει ε, να έχουμε και την απαραίτητη ε, και θα το κάνουμε να έχουμε δηλαδή τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μα για να εξετάσουμε την δική σα πρόταση οδηγία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αύριο θα γίνει η συζήτηση και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία σύμφωνη τοποθέτηση από την πλευρά του Κοινοβουλίου μεταξύ δηλαδή των πολιτικών ομάδων του να έχουμε μία αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή μέσα στον 21ο αιώνα. Όμω ε, ε, θα πρέπει να σα πούμε από τώρα ότι δεν θα κινηθούμε όπως ε, το Συμβούλιο, αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Δηλαδή, χρυσή τομή, ούτω ώστε να έχουν ένα, μια ευρεία επιτυλία σε προσφορές οι καταναλωτέ και από την άλλη πλευρά να χαίρουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων τους. Αυτό είναι ο στόχος τον οποίο θέλουμε να επιτύχουμε από κοινό μεταξύ μας, ε, με, με, με και... Α, Ελπίζουμε πω αυτό θα γίνει, αλλά θα ήθελα να εκφραστώ και πιο συγκεκριμένα ε, σε δύο σημεία τη παρουσίασή σα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την συλλογική ε, αγωγή, το collective redress. Εμείς ακόμα και μετά από την ε, νέα εκλογή μας έχουμε ε, αρκετές επιφυλάξεις γιατί οι δικές μας αρμόδιες υπηρεσίες μας κατέδειξαν πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τελικά να ισχύσουν αμερικανικού αμερικανικές, ε, αμερικανικά πρότυπα στην ευρωπαϊκή αγορά, ούτω ώστε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ούτω ώστε το σημείο αυτό καμπή να μα οδηγήσει σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δυστυχώ, αυτέ οι δύο ε, ε, προτάσει από τη δική σα πλευρά θα εξεταστούμε με πολύ προσεκτικό τρόπο, τουλάχιστον από πλευρά του ΕΛ, γιατί δεν θέλουμε να συμβεί αυτό που συνέβη στην Αμερική, δηλαδή τελικά να μην έχουν αποκτήσει, να μην έχουν καταφέρει τίποτα οι ίδιοι αλλά να έχουν πλουτίσει τα δικηγορικά γραφεία. Ε, η κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Κούνεβα ε, για την παρουσίασή σας και θα ήθελα να επαναλάβω μία πρόταση την οποία αναφέρατε και είναι κάτι που τη θεωρώ πολύ εύστοχο ότι χρειαζόμαστε δηλαδή μια πολιτική του ενεργού καταναλωτή. Αλλά μια τέτοια πολιτική ενεργού καταναλωτή σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται διαρκώ. Εάν όμω, όπω εσεί προτείνετε, θα πρέπει να υπάρξει πλήρη εναρμόνιση με βάση αυτή την οδηγία, δεν θα ε, διασφαλίζεται ακριβώ αυτή η δυναμικότητα, δηλαδή αυτή η περαιτέρω εξέλιξη και αναπροσαρμογή. Γιατί ακριβώ θα ανακόπτεται η περαιτέρω εξέλιξη ε, μέσω ακριβώς της διαδικασίας και των μηχανισμών που ακολουθούνται κατά την ε, νομοπαραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι τέτοιο δεν το επιθυμούμε. Επιθυμούμε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και όχι για την αγορά, όπως είπε ο κύριος ε, Σουβάμ μόλις τώρα, αλλά για τους ανθρώπους μέσα στην αγορά. Και Γι' αυτό και θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με χαρά μου ε, άκουσα τον ε, κύριο Σεγητή να λέει ότι πράγματι θα ε, αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε στην εξέταση αυτή τη πρόταση, ώστε να μην κάνουμε λάθη εδώ. Το δεύτερο σημείο. Θα είμαι πιο σύντομη. Σε ό,τι αφορά το collective redress, λοιπόν, τι συλλογικέ αγωγέ, συνεχίζουμε να σα υποστηρίζουμε σε ό,τι αφορά την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας. Προφανώς τόσο εσείς όσο και εμείς δεν θέλουμε να ισχύσει ένα αμερικανικό πρότυπο εδώ. Προφανώ. είμαστε η Ευρώπη, έχουμε δηλαδή τη δική μας ε, ε, νομική δομή, δηλαδή τη δική μα νομοθεσία και τελείως διαφορετική νομική συνεργασία μεταξύ μα από ό,τι συμβαίνει στι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι σαφέ. Όμω, εκείνο που θέλουμε εμεί να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ζημιώνονται να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά του και ε, ε, όχι ε, πέρα από τα ουσιαστικά τους, από το ουσιαστικό τους ε, δικαίωμα. Επίσης, εκείνο που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να μεταχειριστούμε ουσιαστικά δυσμενώς, δηλαδή να κάνουμε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ακριβώς θα μπορούν να προσαρμόσουν την τιμολογική τους πολιτική με βάση ε, τα δικαιώματα του καταναλωτή. Άρα λοιπόν θα θέλαμε να σας υποστηρίξουμε σε αυτή την ε, κατεύθυνση των συλλογικών αγωγών και θα συνεχίσουμε να σας ε, στηρίζουμε. Θα εξετάσουμε βέβαια προσεκτικά τόσο όσα όπως είπε και ο συνάδελφος κύριος συζητητής. Αλλά... Και τέλος σε αυτό το γύρο των ερωτήσεων η κυρία Τούρινγκ νέο μέλος, την καλωσορίζουμε κιόλα. Θέλω να μιλήσω δανέζικα. Απλά ενημερώνω τους διερμηνεί Θα θέλαμε... Ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ε, παρουσίασή σας. Ε, θεωρούμε πως η βασική σας προσέγγιση είναι σωστή, δηλαδή πράγματι θέλουμε καλύτερη προστασία του καταναλωτή στην Ευρώπη. Αυτό είναι αδεφισβήτητο, αλλά βέβαια το ερώτημα είναι το πώς θα επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πώς αξιολογούμε το σημερινό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή ε, και τελικά θέλουμε να έχουμε προστασία εναρμονισμένη γιατί όπως ξέρετε είμαστε πολύ επικριτικοί απέναντι σε έναν οργανισμό στο ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Δύο σημεία θα ήθελα να θίξω πιο συγκεκριμένα. Ε, ποια, τι έχετε να μας πείτε σε σχέση με το γεγονός ότι η Επιτροπή ε, στη δική της πρόταση δεν αναφέρει, δεν κάνει μεγάλο λόγο για τα πρότυπα. Ε, έχουμε ακούσει πολλά περί συγκριτικών μελετών, αλλά δεν βλέπουμε πολλά μέσα στην ίδια πρόταση. Οπότε θα μπορούσατε να μα πούτε τι συμβαίνει εδώ. Υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο συνεχίζεται, δηλαδή εργασίε, μελέτε, τι οποίε εκπολείται ακόμα. Ένα ακόμα σημείο. Πολλοί ε, νομικοί από τις διάφορες ε, και δικηγόροι από τις διάφορες ενώσει ε, προστασία των καταναλωτών δεν αντιλαμβάνονται ακριβώ τι προτείνουμε. Άρα λοιπόν δεν αποτελεί μία από τι αρετέ τη νομοθεσία το να γίνεται αντιληπτή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη τη Δανία ε, χρειάστηκε περίπου, χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο για να συντάξει μια δική του έκθεση. Και βασικά αυτό το Υπουργείο κινείται με, εργάζεται γρήγορα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια, μια πρόταση συγγνώμη, η οποία να είναι διαφανή και να αντιλαμβανόμαστε ακριβώ τι προτείνει. Επίτροπε, σας δίνω το λόγο για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε αύριο μία ακρόαση και φυσικά θα συνεργαστούμε, αυτό είναι σαφές. θέλω να κατοχυρώσουμε το βέλτιστο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Θα προσπαθήσω να σας καθησυχάσω. Μπορούμε να πάρουμε τα καλύτερα στοιχεία που έχει κάθε χώρα, αλλά άμα πάρουμε όλα αυτά τα καλύτερα κομμάτια, δεν είμαι σίγουρη ότι, παραδείγματος χάρη, έτσι για να μιλάμε συγκεκριμένα, ε, μέσα επανόρθωσης ε, ζημιών από ένα κράτος μέλος. Ε, νομίζω ότι άμα πάρουμε όλα αυτά τα στοιχεία, αντί να φτιάξουμε ένα καλό παζλ, θα φτιάξουμε ένα Φραγκεστάιν. Γιατί δεν θα υπάρχει συνέπεια, συνέχεια ανάμεσα στα στοιχεία. Οι καταναλωτές, ναι, εμείς δημιουργούμε 58% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλει οδηγία να το αναγνωρίζει σε αυτή την περίοδο της οικονομικής ύφεση, ε, το θέμα είναι πώς θα αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ε, ο καλύτερος τρόπος, κατά τη γνώμη μου, είναι να ε, έχουμε καλύτερα δικαιώματα και το επιτυγχάνουμε αυτό μέσα από την οδηγία. Υπάρχουν δύο συμπληρωματικοί πίνακες που αύριο θα συζητηθούν. Πρώτον, πρόταση οδηγίας για την προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών και επίπτωση σε εθνικό επίπεδο αυτού και σχέση με τους γενικότερους κανόνες για το δίκαιο των συμβάσεων και άλλα κομμάτια της κοινοτική νομοθεσίας. Αυτό είναι ο ένας πίνακας και ο άλλος πίνακας ε, φέρει επί της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και επίπτωση στο εθνικό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Δηλαδή κάναμε αντιπαραβολή κατάρθωση άρθρο για να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος πώς αλλάζει η προστασία, ε, ένα χρόνο λιγότερο παραδείγματο χάρη, 14 ε, ημέρες, αυτό είναι εύκολο να το παρακολουθήσετε τον πίνακα. Ε, στις περισσότερες χώρες έχουμε 14 μέρες, σε άλλες 10. Μόνο σε δύο έχουμε 15 ημέρες μειώνεται η προστασία, μπορεί κατά μία μέρα, αλλά είναι πολύ πιο αξιόπιστο το σύστημα αν υπάρχουν ομοιόμορφοι κανόνες. Φιστώ την προσοχή σας στο θέμα του collective redress, ε, συλλογικής αποζημίωσης. Κατάλαβα τι μου είπατε για τις συλλογικές ε, μηνύσεις ε, στη ΣΥΠΑ. Έχω πει επανειλημμένα ότι δεν μιλάμε για τέτοιο σύστημα συλλογικών μηνύσεων. Έχουμε ρήτρε διασφάλιση, έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχουμε πέντε εναλλακτικέ λύσεις που πόρο απέχουν από τις συλλογικέ μηνύσει. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, αλλά θα σας μιλήσω για τη διαδικασία, γιατί θέλω όλοι να συνεργαστούν στενά μαζί μας για να διαπιστώσετε τη σοβαρότητά μας. στι 27 Νοεμβρίου εξέδωσε πράσινη βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις πιθανές εναλλακτικέ λύσεις για την συλλογική αποζημίωση. Πάνω από 190 απαντήσεις πήραμε από τα κράτη-μέλη, από ενό επιχειρήσεων, νομικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Μετά, για να ενισχύσουμε περαιτέρω το διάλογο με του κοινωνικού εταίρου, κάναμε και τρει διαβουλεύσεις για δύο εβδομάδες, έτσι, και δημόσιες ακροάσεις και, και η, η, συνεχίζεται η διαδικασία. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ προετοιμάζει τώρα μελέτη αντικτύπου όπου εξετάζονται με πάσα σοβαρότητα όλες οι εναλλακτικέ λύσεις. Ε, ε, το Συμβούλιο Αξιολόγηση στις 21 Οκτωβρίου του 2009 θα εξετάζει την πρόταση, δηλαδή Λίαν Συντόμως. Δεν βιαζόμαστε βέβαια σπέβδουμε βραδέως και προφυλασσόμεθα ούτως ώστε να έχουμε στη, ε, περισσότερα εργαλεία που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι καταναλωτές ούτως ώστε να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους. Ε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στη δημοκρατία, ε, ε, καλύτερο από το δικαστήριο, αν πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό για την επανόρθωση της ζημιάς. Εάν ε, αξιώνεται 5 ευρώ, 5 ευρώ θα πάρετε, όχι 6, αυτή είναι η αρχή. Τώρα το άλλο ερώτημα που μου θέσατε για την... Ε, για την απίσχυνση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία. Μα όχι, η οδηγία τα βελτιώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλούς τομείς, αν συγκρίνουμε με την υφιστάμενη νομοθεσία σε διάφορα κράτη-μέλη και απευθύνομαι την ε, τρίτη ομιλήτρια από τη Δανία. Θα σας ε, παραθέσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Με την ε, νέα οδηγία έχουμε καλύτερη προστασία για την απόσυρση, το δικαίωμα απόσυρση των καταναλωτών από μια αγορά, παραδείγματο χάρη. Και αυτό δεν προϋποθέτει επίσκεψη από τον εμπορό. Ε, επίσης, ο καταναλωτής ε, δεν επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος, εκτός αν νωρίτερα έχει ενημερωθεί σχετικά. Επίσης, μιλήσαμε για την περίοδο 14 ημερών. Η πλήρης εναρμόνιση σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν κάπως τους κανόνες τους. Αλλά είμαι πεπισμένη ότι το επίπεδο προστασίας είναι βέλτιστο μέσα στην οδηγία. Σε πολλές ε, περιπτώσεις έχουμε αυστηρότερους κανόνες ε, μέσα ε, σε κάποια νομοθετικά κείμενα, αλλά στην ουσία αυτό δεν συνεπάγεται καλύτερη προστασία στην πράξη. Παραδείγματο χάρη, νομικό, νομική εγγύηση για πάνω από δύο χρόνια. Πώς θα αποδείξει ο καταναλωτή ότι αυτά τα προϊόντα ήταν ελαττωματικά ήδη από την αρχή άμα έχει περάσει τόσο καιρό. Και Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά πριν ακούσω τις επόμενες ερωτήσεις θέλω να σας πω ότι πάτε στη διάθεσή σας είμαι. Απλά ε, ειδοποιήστε με ότι θέλετε να μου μιλήσετε Ειδοποιήστε τους συνεργάτες μου και με μεγάλη χαρά θα έρθω και θα συζητήσω με ε, οποιοδήποτε μέλος Επιτροπής εκδηλώσει ενδιαφέρον στη, ε, στη δουλειά μου. Μα όλοι ενδιαφέρονται. Ξέρετε πώς έχουμε στον κατάλογο των ομιλητών λέει ο κύριος Χάρμπορ, και συνεχίζει και μεγαλώνει ο κατάλογος. Όχι, μας ενδιαφέρουν αυτά που λέτε και αναφερθήκατε σε κάποια έγγραφα τα οποία θα είναι όντω διαθέσιμα και θα κάνουμε πλήρη συζήτηση και αύριο. Έχετε το, το κατά νου, συνάδελφοι, στι ερωτήσει σας. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τι τρει επόμενε. Η κυρία Σάλντε Μόσα, ο, κύριο ο κύριος Ρίπχολτ και ο κύριος Γοσφό. Πρόεδρε, εσείς είστε τρίτος, κύριε Γοσφό. Κύριε Σάλντε Μόζε, Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο για την τόσο καλή παρουσίασή της. Ε, σίγουρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι εδώ στόχος είναι η βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων τη ε, εσωτερική αγορά Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ε, μπορούν να βελτιωθούν οι κανόνες αυτοί. Για παράδειγμα, είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου αγόρασε ένα ταξιδιωτικό πακέτο ε, ο καταναλωτής ε, από μια εταιρεία που δεν είχε έδρα ε, στο κράτος διαμονής, οπότε οι εθνικές αρχές πολύ δύσκολα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το όλο ζήτημα σε περίπτωση που είχαν προβλήματα κτλ. Επίσης, οι αγορές μέσω του διαδικτύου. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο να εγγυηθούμε πρακτικά ε, την, ε, ε, τα, ε, ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτά τα θέματα πρέπει να συστηθούν στις λεπτομέρειές τους. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το γενικό έβρος της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στη χώρα μου, στη Δανία. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα για το τι θα συμβεί Ω αποτέλεσμα τη οδηγία αυτή Τι θα συμβεί σε σχέση με το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Γιατί εξακολουθεί να λείπει μία μελέτη συγκεκριμένη των πρακτικών συνεπειών σε επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση βεβαίω που, αρχίσει, που τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθεσία. Εμείς, σα λέω, με βάση την νομοθεσία τη χώρα μα, ζητήσαμε να γίνει αυτή η μελέτη πριν από ένα χρόνο και όμως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το ζήτημα στι λεπτομέρειέ του και σίγουρα θα το συζητήσουμε και αύριο. Πάντω ήθελα να μου το σχολιάσετε και στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή. Ο κύριο Ρέπο. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, έχω μία πρακτική φύσεως ερώτηση. όσον αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς στις σκανδιναβικές χώρες. Ε, σε σχέση με τα, γρήγορα δάνεια. Ε, και αυτό το φαινόμενο εξαπλώνεται και με ιδιαίτερη ταχύτητα και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, μπορεί κανείς να δανειστεί μικρά χρηματικά ποσά, βεβιασμένα θα έλεγα. Βιαστικά. και το επιτόκιο υπολογίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενό μηνό. Από το διαδίκτυο κανεί μπορεί να πάρει τα δάνεια αυτά. Αυτό καλύπτεται από μια νέα οδηγία για τους καταναλωτές. Αλλά επειδή τα ποσά είναι μικρότερα από τα 200 ευρώ, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα το ποια νομοθεσία εφαρμόζεται. Άρα, το επιτόκιο, το ετήσια υπολογιζόμενο επιτόκιο, ε, σε ορισμένε περιπτώσει είναι πάνω από 200, άλλε φορέ δεν πάνω από το 1000%. Για να σα πω την αλήθεια, ο μέσο όρο είναι 500%. Τι γίνεται λοιπόν, οι, ε, πολλές φορές οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, ε, προβλήματα ε, ε, ε ή ε, χαρτοπεξίας, είναι πολύ εύκολο με τον τρόπο αυτό να μπουν σε αυτό το φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης. Σα... Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή. Έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία για το ζήτημα αυτό και έχετε την πρόθεση να αναλάβετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για να ε, ρυθμίσουμε και τον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Ε, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, σας ενημερώνω και ήταν πολύ συνάδελφοι εκεί πέρα. Ο κύριος Ροσφόρ επιτέλους, ναι αυτή τη φορά είναι η σειρά μου. Ε, Επίτροπε, θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι αναγνωρίζουν την αξία της δουλειάς σας ε, ήδη και στην προηγούμενη θητεία. Ελπίζω να σας δοθεί ευκαιρία να συνεχίσετε πρέπει να εξελίσσονται τα δικαιώματα όπως και η ίδια η κατανάλωση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, το βλέπουμε παντού. Ε, παραδοσιακά ε, πουλούσαμε απλά πράγματα, τώρα πουλάμε πακέτα, υπηρεσίες, όλα επιγραμμικά. Χρειάζεται εναρμόνιση και ένα πράγμα ε, που εκτιμώ πραγματικά στο πρόγραμμα σας είναι το εξή. Η ενημέρωση είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή. Ό,τι και αν πει κανείς, διαφέρουν τα δικαιώματα από χώρα σε χώρα, αλλά ε, το κοινό σημείο είναι ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του, γιατί τα δικαιώματα αυτά είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Ε, εάν μέσω της εναρμόνισης μπορούμε επιτέλους να διασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής ε, θα γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά του, αυτό καθεαυτό συνιστά μεγάλη πρόοδο. Κάτι άλλο που, στο οποίο αναφερθήκατε, για την εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές. Κατά τη γνώμη μου ε, δεν αντιτίθεται αυτό στη δυναμική πορεία των επιχειρήσεων. Ε, είναι αλληλοσυμπληρούμενα αυτά τα στοιχεία. Αλλά πώς να εξασφαλίσουμε διαφύλαξη ή βελτίωση των δικαιωμάτων γνωρίζοντας ότι ε, στις χώρες μας και δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στη Γαλλία, αν είμαστε πιο εξελιγμένοι ή όχι, δεν έχει και σημασία. Αλλά παντός αν η εναρμόνιση οδηγεί σε υποχώρηση, πώς ακριβώς θα πουλήσουμε αυτό το πακέτο στου πώς θα παρουσιάσουμε μια Ευρώπη που για ένα σημείο που, που δεν φαίνεται τόσο σημαντικό ε, όσο τα υπόλοιπα, πώς θα παρουσιάσουμε λοιπόν ένα πακέτο που συνιστά υποχώρηση, δηλαδή χρειαζόμαστε στοχευμένη εναρμόνιση. Μήπως αυτό είναι μια ιδέα που θα έπρεπε να αναπτύξουμε περαιτέρω σας ε, συγχαίρω για αυτά που κάνατε για τα ε, τραπεζικά έξοδα την περασμένη εβδομάδα. Είναι πολύ θετικό, απλά θα θέλαμε να αλλάξουν τα πράγματα ε, στα κράτη-μέλη μετά από αυτή την πρωτοβουλία σας και πώς θα συντονίσετε τη δράση σας, τη δράση της συναδέλφου σας, της κυρίας Νέλη Δηλαδή, μέσα στην ίδια επιτροπή δεν θα έπρεπε να έχουμε δύο διαφορετικά μηνύματα. Θα χρειάζεται κοινή προσέγγιση. Κύριε Ροσφόρ, σας ευχαριστούμε και ξέχασα να σας καλωσορίσω και εσά στην Επιτροπή. Καλωσορίσατε. Ήταν η πρώτη σας παρέμβαση εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω στους ε, φίλους από τη Δανία ότι πράγματι το επίπεδο προστασίας στη Δανία είναι πολύ ψηλό. Και αυτό είναι καλό. Και μπορούμε βεβαίως να ακολουθήσουμε όλα αυτά τα καλά παραδείγματα που ε, δίνουν αυτές οι οργανώσεις των καταναλωτών που έχουν ε, ιστορία 60 ετών και που έχουν, ε, είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην προστασία των καταναλωτών. Αλλά κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Η κάθε χώρα πιστεύει ότι είναι η καλύτερη στο θέμα τη προστασία των καταναλωτών. Ή σχεδόν κάθε χώρα. Ακριβώ γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε και να δούμε. Και κοιτάξτε, η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη. Θέλετε να συνεργαστούμε για το καλό του Ευρωπαίου καταναλωτή. Και πώς θα το κάνουμε εάν ο καθένας οχυρώνεται ε, στις εθνικές του θέσεις, εθνική προστασία της εθνικής αγοράς. Μπορείτε να εξηγήσετε στους καταναλωτές μας σήμερα που αγοράζουν προϊόντα online. Κοιτάξτε, ε, το κατάστημα πλέον είναι η οθόνη, ούτε καν το υπολογιστή του κινητού σας. Εγώ δηλαδή ως δανός καταναλωτής προστατεύομαι ε, με τον καλύτερο τρόπο. Μα δεν είναι αλήθεια. Αυτό ισχύει μόνο αν ψωνίζετε μόνο εντός των εθνικών σας συνόρων. Αυτό όμως σημαίνει πρώτα απ' όλα δεν έχετε αρκετές επιλογές και δεύτερον αντιμετωπίζεται λιγότερο ανταγωνισμό στην αγορά. Ακόμα και για του ε, παραγωγού παραγωγούς ε, και πάροχου προϊόντων και υπηρεσιών. Πρέπει να ανταγωνιστούν του υπόλοιπου και να μπορούν να συγκρίνουν. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το διαδίκτυο, δεν μπορούμε να το κλείσουμε και να το περιορίσουμε στα σύνορα κάθε εθνική αγορά. Γι' αυτό σα παρακαλώ, κοιτάξτε τον πίνακα σύγκριση, το συγκριτικό πίνακα που πήρατε. Και εκεί θα, θα δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες με ακρίβεια. για τα επιμέρους εθνικά ζητήματα. Αλλά θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι σε κάθε σημείο του κειμένου θα βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών στην Δανία. Γιατί εδώ πρέπει να δούμε και τη σχέση κόστος-οφέλους. Αυτό μα ενδιαφέρει κυρίω όταν καταρτίζουμε νομοθεσία. Μιλάμε για καταναλωτέ. Εγώ εσκεμμένα ακολουθώ αυτή την, προσ... την προσέγγιση. Αλλά δεν ξεχνώ και τι επιχειρήσει. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, όταν. Ε, όταν μειώνουμε τη γραφειοκρατία κατά 97% με αυτή την νομοθεσία, μα θα ωφεληθούν και επιχειρήσει. Θέλουμε να αυξήσουμε του ρυθμού ανάπτυξη. και έχουμε διασυνοριακό εμπόριο 8 ή 9%. Με τη βεβαιότητα και με την εμπιστοσύνη. Αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά 2, 3, 5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στα επόμενα χρόνια. Μα αυτό θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση της αγοράς. Βεβαίως καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Και σας παρακαλώ κοιτάξτε με προσοχή τον πίνακα. Η Επιτροπή συνήθως δεν είναι υποχρεωμένη να δίνει το συγκριτικό αυτό πίνακα το Συμβούλιο κάνει τις συγκρίσεις και δίνει τις σωστές απαντήσεις. Αλλά όπως σας είπα και εγώ και οι συνεργάτες μου, θέλουμε, επιθυμούμε να σας δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες, περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες σύγκρισης. Λοιπόν, όσον αφορά ε, αυτά τα δάνεια, πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Πριν από δύο χρόνια είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Όταν είχαμε προκηρύξει ένα διαγωνισμό για τα καλύτερα ε, σχέδια συνειδητοποίηση των καταναλωτών και ε, κέρδισε το βραβείο ο Δανικός, ο, Δανικός Οργανισμός Προστασίας των Καταναλωτών όσον αφορά αυτά τα δάνεια μέσω ε, των κινητών τηλεφώνων ε, και των μηνυμάτων σε σχέση με τις καλύτερες πρακτικές. Τώρα, όσον αφορά τα δάνεια αυτά τα οποία προσφέρονται μέσω των κινητών τηλεφώνων και των μηνυμάτων, είναι μια πρακτική στη Φινλανδία, Σουηδία, στην Εστονία ε, και τώρα ε, διαδίδεται και σε άλλε χώρε τη Βαλτική, Δημοκρατία τη Βαλτική. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν το εξή, ότι σε παρόμοιε περιπτώσει και οι προποθέσει τη οδηγία για την καταναλωτική πίστη και ε, η ε, παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεων, αποστάσεως ισχύει. Α εφαρμόσουμε λοιπόν νομοθεσία, νομίζω ότι αρκεί. Κύριε Ρόσφορ, και εγώ ε, θα ήθελα να σας πω ότι είναι εξαιρετικό το βιβλίο σας για τους καταναλωτές. Να ανταποδώσω την φιλοφρόνηση. Πάντως, να πω το εξής. Όσον αφορά την ευκαιρία που ε, μας δίδεται να δούμε από τη μια ε, τα συμφέροντα των καταναλωτών και από την άλλη το κόστος της επιχειρήσης. Μα κοιτάξτε, αυτό πρέπει, αυτά πρέπει να τα βάλουμε στην πλάστικα. Και όπως είπατε κι εσείς, μόνο εάν υπάρχουν κοινοί κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ε, συνειδητοποίηση των καταναλωτών. Ε, για την, ε, γιατί διαφορετικά τι να κάνει η Επιτροπή, να εξηγεί τα δικαιώματα στη Φιλανδία, στη Γαλλία, στη Δανία σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσα να παραβιάσω και τις αρχές της επικουρικότητας. Όσον αφορά τη συλλογική αποζημίωση. Εδώ να ξεκαθαρίσω το εξή. Εμείς το βλέπουμε το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Εκεί ασχολούνται με την ε, νομοθεσία αντιτράστ ε, και από τη σκοπιά των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως πιθανά θύματα. Εμείς όμως ασχολούμεθα με το θέμα της αποζημίωσης. Όταν κάποιος χάνει κάτι, πρέπει να πάρει τα ίδια χρήματα που έχασε. Και αυτό να γίνει συλλογικά. Το, το, ακριβώς το ίδιο χρηματικό ποσό. Αν δεν με βοηθήσετε να σας εξηγήσω σε τι θα ωφεληθούν ε, οι καταναλωτές, στη Γαλλία για παράδειγμα, να εξηγήσω στη Γαλλία, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι ε, να βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν θα υπάρξει μια κοινή αγορά ε, των πολιτών και των καταναλωτών. Σας ευχαριστούμε. Ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο, οπότε ε, ζητώ από την επόμενη ομάδα ομιλητών να είναι εξαιρετικά σύντομη και σαφής. Η κυρία Κανιέτη, ο, ο κύριος Τεραμπέλα και η κυρία Ράπτη. Κυρία Κανιέτη, παρακαλώ. Και παρεπιπτόντας να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω λετωνικά. Θα ε, δράτω με της ευκαιρίας για να σας ευχαριστήσω, Επίτροπε. Ήταν σαφέστατη η παρουσίασή σας. Θα θίξω δύο εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα. Είμαι νέο μέλος της Επιτροπής και θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση στην Λετωνία. Συχνά έρχομαι σε επαφή με οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών και εκπροσώπους των επιχειρήσεων και ε, κρίνω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει σύγκληση απόψεων και να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Όλοι πιστεύουν ότι έχουν δίκιο και μένουν στη θέση τους. Ποια θα είναι αυτή η κοινή γραμμή, πώς ακριβώς θα υπάρξει σύγκληση αυτών των ε, αντίστοιχων απόψεων. Η Λετωνία διέρχεται μια σοβαρή οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή. και θεωρείται πολυτέλεια, είδος πολυτέλειας να υπάρχουν οργανισμοί προστασίας των καταναλωτών και το κονδύλι μας έχει μειωθεί κατά 30%. Δεν υπάρχει μη καπαόμικρον για την προστασία των καταναλωτών στη Λετωνία. Υπάρχει μόνο ένα κέντρο προστασίας των καταναλωτών. Αν μειωθεί το δυναμικό του λοιπόν, λόγω της περικοπής των κονδυλίων, κανείς δεν θα γνωρίζει καθόλου τα, ποια είναι τα δικαιώματά του ως καταναλωτής. Μπορείτε να μας ενημερώσετε ακριβώς πώς ε, θα προωθήσετε την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χρειάζεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε χώρες όπως η δική μου, κυρίως σε περιόδους κρίσης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τεραμπέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Λέγατε πριν ότι ο καταναλωτής και ο πολίτης πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ενιαία αγορά, να τον υιοθετήσουν. Μα δεν μπορούν αν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δείχνουν μέσα από μελέτες ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες, ανακολουθίες και δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα. Ε, όπως είπε και ο κύριος Γοσφό, ε, ε, την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τα ε, ε, τραπεζικά τέλη. Ε, πριν από 20 χρόνια ο Κάλφαν Μίρτε, πρώτος αρμόδιος επίτροπος, είχε κάνει μια αντίστοιχη μελέτη που είχε καταλήξει στα ίδια πορίσματα. Τι έγινε στα ενδιάμεσα 20 χρόνια, χιλιάδες μελέτες. Αλλά, ωραίο, καλό και αυτό. Αλλά κάνοντας μελέτες δημιουργείται μια επιθυμία στον καταναλωτή ότι κάτι θα αλλάξει σε σχέση με αυτή την δυσπραγία. Τα κράτη-μέλη φυσικά πρέπει να υπομισθούν τις δικές τους ευθύνες γιατί υπάρχουν και εθνικοί κανόνε. Εγώ θα πάρω ένα παράδειγμα. Θα μιλήσουμε για τους καταναλωτέ και όχι για νομοθετικές διατάξεις. Ε, το, το, το roaming η περιαγωγή παραδείγματο χάρη. Αυτό μας επηρεάζει όλους. Ε, είναι εντελώς αδιαφανές το σύστημα ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπερηφανεύεται ότι ρύθμισε το πρόβλημα. Όπως και σε άλλους τομείς, ε, επίτροπε, ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας γιατί μετά από τις μελέτες που τις πληρώνει ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος πρέπει κάτι να κάνουμε για να λύνουμε και το πρόβλημα. Μόνο έτσι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών γιατί ε, σωστά διαπιστώσατε ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα μέσα από τις μελέτες ε, που ε, κάνετε. Κυρία Ράπτη τώρα. Κυρία Κούνεβα, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω εδώ. Παρακολουθώ με πολύ προσοχή τη δουλειά σας. Προέρχομαι από την Ελλάδα όπου έχουμε προβλήματα. Μιλήσατε προηγουμένως και είπατε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, ούτε οι έμποροι ε, θα προσθέσω εγώ, ε, μερικές φορές όμως τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι τράπεζες, αλλά κάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των τραπεζών ή όχι. Ε, πριν από αρκετούς μήνες στην Ελλάδα 17 τράπεζες πλήρωσαν πρόστιμο γύρω στα 10 δις ευρώ και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ωστόσο η κακή πρακτική συνεχίζει. Και επειδή μπροστά μας δεν έχουμε μόνο το παρόν αλλά έχουμε και το μέλλον και επειδή ήδη έχει, έχουμε προχωρήσει στον ορισμό του κυρίου Μπαρόζο στην επόμενη Επιτροπή, ε, βλέπω ότι υπάρχει μία ε, διάσταση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ανάμεσα σε αυτό που απήντησε ο κύριος Μπαρόζο όταν ήρθε στη σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου και στην οποία είπε πάρα πολύ απλά ότι κοιτάξτε να δείτε οι αρχές των κρατών μελών δεν είναι συνεργάσιμες. Απ' την άλλη πλευρά διάβασα με πάρα πολύ προσοχή ένα απόσπασμα ομιλία σας στις 22 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το οποίο το λέω επιλέξει λέτε και πάρα πολύ σωστά ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια συνολική προσέγγιση που θα αναπτύσσει ένα πλαίσιο σχετικά με συγκεκριμένα στάνταρς, σχετικά με την ενημέρωση των πελατών, τα οποία θα πρέπει να γίνονται ε, σεβαστά από τους Συμβούλους Τραπεζικών Υπηρεσιών και τα οποία θα πρέπει να επιβάλλονται από όλες τις αρμόδιες αρχές. Και σας ρωτώ ευθέως, πόσο αισιόδοξοι είστε ότι η νέα Επιτροπή θα μπορέσει μετά και από αυτά που δήλωσε ο κύριος Μπαρόζο σε εμά να το κάνει αυτό πράξη. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ναι, νομίζω πως ε, θα είναι δύσκολο να καταλήξω εδώ τη συζήτηση γιατί οι ερωτήσεις γίνονται ολοένα και πιο ενδιαφέρουσες ε, ε, και πιο προσφυγεί για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ε, κύριε Γανιέτη, σε ό,τι αφορά ενημερωτικέ εκστρατείε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ναι, αυτέ θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στην Ευρώπη σε επίπεδο κρατών μελών, εάν υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα. Σε διαφορετική περίπτωση, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει πιο συγκεκριμένα στις νέες ε, χώρες, νέα, 12 νέα κράτη-μέλη, όπως γνωρίζετε ήδη χρηματοδοτεί ε, τέτοιες ε, δράσεις ε, όπου την κύρια συγχρηματοδότηση, το κύριο μερίδιο το χρηματοδότηση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω καλά την κατάσταση στη δική σας χώρα γιατί την έχω επισκεφθεί και έχω συνομιλήσει με τις δικές σας ενώσεις προστασίας των κανοντών και συνεργαζόμαστε με την ΠΕΟΥ ούτως ώστε να επιτύχουμε μια πιο ομοιογενή προσέγγιση και να ενδυναμώσουμε τις ενώσεις των καταναλωτών. Αντιλαμβανόμαστε πως αποτελεί πρόβλημα αυτή η κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμεί περισσότερη βούληση μεταξύ των ενώσεων προστασία των καταναλωτών για να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ του, αλλά δεν θα ε, σταματήσουμε να μεταβαίνουμε εκεί, να προσπαθούμε και ε, θα προσκαλέσουμε τι ε, ενώσει προστασία των καταναλωτών κατά τη διάρκεια του συνεδριάσεων του να προσπαθήσουν να βοηθήσουν την κατάσταση στη χώρα σας. Νομίζω πως δεν πρόκειται για πολυτέλεια. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πολυτέλεια το να βόμαστε τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ε, το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Όταν δηλαδή η καιρή είναι δύσκολη, όταν η πιστοσύνη πίστη στην αγορά πλήττεται, χρειάζεται ακριβώς να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στην αγορά. Ε, και γι' αυτό ζητώ από τις κυβερνήσεις μας να συνεισφέρουν περισσότερο χρηματοδοτικά. Και να κλείσω αυτό το σημείο λέγοντας ε, πως με αυτό το scoreboard, το European Market Scoreboard, θα, μπορούσε, θα μπορούμε στο τέλος να συγκρίνουμε τα ποσά που αφιερώνουν τα κράτη-μέλη στις δική τους ε, πολιτική προστασία του καταναλωτή. Γιατί δεν πρόκειται ε, ε, για ε, χρήματα πεταμένα δηλαδή, θα μπορούσαμε να, ε, έχουμε και τις, ε, τους επιθετές που έχουμε τόσο πολλούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να α, τους θεωρήσουμε ως μια επένδυση την οποία κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τέτοιου είδου στοιχεία στην διάθεσή μας στο μέλλον. Θα μπορέσουμε, λέγοντάς το ανοιχτά, να ασκήσουμε περισσότερε πιέσει στι εθνικέ κυβερνήσει. Είχα λοιπόν τη δυνατότητα να συναντήσω τον κύριο Γκάρμπαν ε, και βέβαια είχα την, την τιμή να γνωρίσω έναν άνθρωπο του οποίου το όνομα συνδέεται με, με το προσθέσεις του καταναλωτών τόσο πολύ. Απαντώντα λοιπόν στο ερώτημά σα, ναι, πράγματι αυτό ο τομέα αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και υποχρέωση για εμά, με βάση τα όσα προβλέπει η συνθήκη. Και ταυτόχρονα η επιβολή του νόμου, το law enforcement, δεν σταματάει στα εθνικά σύνορα και για να επιτευχθεί διασυνοριακά χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και είμαστε διατεθειμένοι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, βοηθήσουμε ούτως ώστε να ενοριακά επιβολή και να υπάρχει περισσότερη συνεργασία στον χώρο της επιβολής. Ακόμα και τώρα όταν συζητάμε το ζήτημα των regulators, αυτή, ε, μια τέτοια απόφαση θα ήταν πολύ χρήσιμη. Γιατί ακριβώς θα μπορούσαμε να δώσουμε περιεχόμενο τελικά στο τι θα κάνουν αυτοί οι regulators. Για παράδειγμα, σε σύγκρουση συμφερόντων αυτό είναι παράδειγμα από γερμανική μελέτη, έτσι, αμυγός γερμανική μελέτη. Είχαμε λοιπόν έναν αγοραστή, ε, μια χείρα υποτιθέμενη, η οποία ε, μετέβησε 25 ε, τράπεζες και σε 24 δεν έλαβε καλές συμβουλές. Και γιατί? γιατί ο μισθό, ε, τον οποίο θα λάβει το εν λόγω άτομο το, ε, ε, το οποίο εργάζεται για λογαριασμό της τράπεζας εξαρτάται και από την τιμή του προϊόντος το οποίο θα απολύσει. Άρα λοιπόν έχουμε μια ευκαιρία εδώ να λάβουμε δράση νομοθετικά και αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει στα ελληνικά, Επίτροπο στην κυρία Ράπτη, για την αναφορά που κάνατε ε, σε αυτές τις 17 τράπεζες ε, και νομίζω πως η Ιταλία έχει κάνει εδώ πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά ε, τα ringtones σε σχέση και με την δική της αρχή ανταγωνισμού και είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα αποτελέσματα της αγοράς για τους καταναλωτές μέσω αυτών των ελέγχων sweeps ε, θα έχουμε λοιπόν αποτελέσματα και από εκεί και σε ό,τι αφορά τι αθέμητε εμπορικέ ε, πρακτικέ και στον χρόνο των τραπεζών. Εμεί συναντηθήκαμε με του εκπροσώπου τη Δυτική ε, Ένωση Τραπεζών και πριν από 1,5 χρόνο περίπου και ήδη είχαμε ακριβώς τέτοιου είδους ανησυχητικά ανησυχίες ενδείξεις σε ό,τι αφορά δηλαδή πωλήσει με άσκηση πίεσης ε, στον ε, καταναλωτή. Ήδη προετοιμάζουμε κάτι εδώ και ακριβώς θα πρέπει να ε, μείνουμε στα αυτά τα οποία συμφωνήσαμε εμείς από κοινού μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 7 ακόμα μιλητέ. Σε ομάδες των τριών πάλι, αλλά σας παρακαλώ πολύ να έσαστε ε, σύντομη. Σε ένα... Ρωτάτε σύντομα. κυρία Στήρα λοιπόν θα αρχίσει, ο κύριος Μίλαν στη συνέχεια και στη συνέχεια η κυρία Βάιλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Όσον αφορά την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, καταλαβαίνω πολύ καλά τα επιχειρήματά σας για την αρμόνιση. Αλλά εδώ υπάρχουν φόβοι ε, όσον αφορά, για παράδειγμα, τη δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με το 15, άμα μειωθεί μπορεί να αισθανθούν ορισμένοι ότι μειώνεται η δυνατότητά τους. Ακόμα και σήμερα το πρωί, ε, στα, στα νέα το πρωί, ε, ακούστηκε ότι ο Μάρκ Σπένσερ είχε στην αρχή 90 ημέρες δοκιμαστική περίοδο, τώρα έγινε 45. Καταλαβαίνετε ε, δηλαδή, παρόλο που και ακόμα το, το χρονικό διάστημα αυτό είναι πολύ μεγάλο, όταν κανείς βλέπει να μειώνεται, να μειώνεται τα δικαιώματά του, ε, αγανακτά. Ε, και κάτι άλλο, όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή ε, και το θέμα της επιβολής των αποφάσεων και κυρίως ε, το θέμα των οδηγών των πόλεων. Πάλι παίρνουμε ανισχυτικά ε, μηνύματα από τους καταναλωτές ε, και για το, για γεγονός ότι παραπλανήθηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και θα πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις ήταν. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω τα πολωνικά. Σας ευχαριστούμε ε, κύριε Επίτροπε για το έργο σας και ε, είμαι σίγουρη ότι θα εξακολουθήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί ασχοληθήκατε με το αμφιλεγόμενο ζήτημα της διαφήμισης ε, και της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Μην ξεχνάμε όλοι ότι Κοιτάξτε, όλα αυτά στηρίζονται στη συλλογή ε, πληροφοριών για τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Και πολλέ φορέ τα στοιχεία συλλέγονται χωρί συγκατάθεση των ενδιαφερομένων. Ε, χρησιμοποιούν λοιπόν πολλοί αυτή την τεχνική, αλλά πολλοί θεωρούν ότι αυτό αποτελεί παραβίαση του ιδιωτικού απορρίτου. Ε, ιδιαίτερα το θέμα του απορρίτου ε, τη αλληλογραφία και τη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, του απορρίτου των προσωπικών δεδομένων. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς βλέπετε το ζήτημα. Ε, ξέρω ότι εσείς προτίθεστε να ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό και να το δείξετε ε, ε, σοβαρά και στις επαφές σας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Γιατί στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς βλέπετε στο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Κρατσαμπίλτ. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε για τις προσπάθειές σας για να, υπάρξουν, ε, για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση, αλλά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για τον καταναλωτή. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν την εσωτερική αγορά. Θα δώσουν ε, και ταυτόχρονα θα δώσουν πολύ υψηλότερο επίπεδο προστασία του καταναλωτή, περισσότερη διαφάνεια και ε, περισσότερο ανταγωνισμό, πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν του πάντε. Κοιτάξτε, Είχαμε εδώ την ε, Σουηδό ε, Υπουργό Αρμόδια για τα θέματα αυτά και τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν στον πιο γρήγορα κοινοί κανόνε. Είπε ότι πιστεύει και βλέπω εδώ ότι ορισμένοι συνάδελφοι έφτιαξαν το ζήτημα αυτό και από τη Δανία και από τη Σουηδία και από τη Γαλλία. Δηλαδή, ε, να διατηρήσουμε υψηλά πρότυπα προστασία του καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και τι ανησυχίε του επιχειρηματικού κόσμου τη Ευρώπη, όπω για παράδειγμα ε, των επιχειρηματιών από τη Γερμανία. Ρωτώ, όταν έρχεσαι σε επαφή με, τον, ε, με του επιχειρηματίε στην Ευρώπη, γνωρίζετε ότι υπάρχουν ορισμένοι που βλέπουν με, με επιφυλακτικότητα τι προτάσει σα. Τι όμως σας λένε συγκεκριμένα και τι απαντάτε εσείς όσον αφορά αυτή τη δυνατότητα εναρμόνισης και αντιστήχησης ε, μιας δυναμικής πορείας των επιχειρήσεων αλλά και, ε, και υψηλού επίπεδου προστασίας των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Λοιπόν, ξεκινώ με την κυρία Στήλερ. Το answer to... Όσον αφορά ε, τις ανησυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς εμάς δεν μας ενδιαφέρει το ζήτημα της εμπορικής εγγύησης. εδώ οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες, είναι, είναι ελεύθερες να ε, κάνουν τις δικές προσφορές. Δεν υπάρχει θέμα. Όσον αφορά τις αεροπορικές ε, εταιρείε. Μετά από ένα χρόνο ε, εργασίας με τις, ε, προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μεγάλη πρόοδο. Δεν θέλω να κατανομάσω, αλλά πρέπει να σας πω ότι λίγες ήταν ε, οι χώρες που επέδειξαν το αρκετό θάρρος έτσι ώστε να κατονομάσουν συγκεκριμένα τις εταιρείε που δεν προστατεύουν τους καταναλωτές. Το αφήνω λοιπόν να το σκεφτούμε για το μέλλον. Εγώ θαυμάζω ιδιαίτερα τις ε, σωστές επιχειρήσεις. Ε, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε ε, με ανθρώπους που ακολουθούν τέτοιες τακτικές, γιατί να μην τους κατανομάσουμε. Ιδιαίτερα λοιπόν όταν έχουμε το διαδίκτυο και όταν το δικό μου παράπονο ως καταναλώτριας μέσω του Facebook, για παράδειγμα, μπορεί να φτάσει παντού. Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ διστάζουμε. Τώρα, όσον αφορά του οδηγού ε, των πόλεων. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μετά από τρία χρόνια προσπαθειών, έγραψα στου ε, ε, αρμόδιου υπουργού, στι οργανώσει των καταναλωτών. Δεν είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με του καταναλωτέ. Αφορούν, ε, είναι, είναι θέμα από, από επιχειρηματία σε επιχειρηματία. Εξακολουθώ όμω να παίρνω παράπονα. Ξέρετε ότι ε, έχουν αναποθέσει τις προσδοκίες τους σε εμά. Μίλησα με την ε, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ε, Αφορών συγγνώμη, δεν κάνω, μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Η συνειδητοποίηση και η ενημέρωση ίσως είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να προσφέρω σε αυτό το στάδιο. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Μπιελάμ, ναι, συμπεριφορά και στοχοθέτηση, να σα πω το εξή στείλαμε μία αποστολή διερευνητική στι Ηνωμένε Πολιτείε την περασμένη εβδομάδα για να μελετήσει το θέμα αυτό. Και ξεκίνησα δημόσια διαβούλευση ε, για ε, την ε, συλλογή προσωπικών δεδομένων και στοιχείων. και, και υπάρχει και ένα φόρουμ. Ένα χρόνο θα συζητήσουμε και στη συνέχεια θα υπάρξει δυνατότητα υποβολή προτάσεων. Σα παρακαλώ λοιπόν, ελάτε με τι απόψει σα. Για την κυρία Μπιλτ και την ερώτησή σα, Πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, οι καταναλωτέ τη Σουηδία ε, ω αποτέλεσμα του CRD θα έχουν περισσότερες, ε, περισσότερη προστασία και περισσότερε καταναλωτικέ προσφορέ, θα έχουν καλύτερο επίπεδο προστασία και πράγματι το CRD, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών βοηθά ιδιαίτερα και θα δώσει και νέο ορμή στι επιχειρήσει. Πώ αντιδρούν ε, οι, επιχειρήσει επιχειρήσεις και ε, αναφερθήκατε στο παράδειγμα τη Σουηδία, μα παντού ισχύουν τα ίδια. Όσον αφορά τη μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου. Τώρα, αν είσαστε μια μικρομεσαία επιχείρηση και μεγάλη, και χρειάζεται 2.157 ευρώ. Όχι, διορθώνει. 257. για να για να καταλάβετε ε, τι γίνεται σε επίπεδο καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Τώρα όμως το ποσό αυτό θα μειωθεί πολύ περισσότερο. Δεν, δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μας πιέζουν για να εγκριθούν οι εθνικοί κανόνες μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής ε, ε, κοινότητας. Αλλά κοιτάξτε, εμείς διαπραγματευόμαστε ε, γενικά. αυτή είναι η απάντηση της συναδέλφου. Ε, διαπραγμάτευση, συζήτηση, μέχρι να υπάρξει συνένεση. Χωρίς όμως τη δική σας συμβολή όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ βοηθήστε μας να, το, να τα πράξουμε όλα αυτά από κοινού. Okay. I think... Uh, θα ακούσουμε τρεις ακόμα μιλητές. Ε, είχαμε τρεις ακόμα μιλητές οι οποίοι ζήτησαν πολύ αργά το λόγο δυστυχώς. Λοιπόν, ο ε, κύριος Κορέα, ο κύριος Μπουζό και ο κύριος Τριανταφυλλίδη και θα κλείσουμε μετά. Ο κύριος Κορέα λοιπόν αρχίζει. Ε, Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για μια πραγματικά εξαιρετική παρουσίαση. Ε, προφανώς και δεν είστε σε θέση να διασκεδάσετε όλες τις ανησυχίες που εκφράζουμε από τη δική μας πλευρά και που εκφράζονται και από την πλευρά πολλών ε, ενώσεων ε, που εκπροσωπούν τους καταναλωτές. Η Επίτροπο μας είπε ότι μπορεί να μας εγγυηθεί ότι τάσεται υπέρ του, των δικών μας στόχων και αυτό δεν το αμφισβητούμε. Προφανώς και το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση της προστασίας του καταναλωτή. Όμως τα επιχειρήματα τα οποία ακούσαμε είναι επιχειρήματα τα οποία ε, στηρίζονται στην φρόνηση αν θέλετε. Δηλαδή ακούμε πάντα το θεωρώ, το φρονώ, το πιστεύω πώς. Ε, θα λάβουμε έναν ε, συγκριτικό πίνακα εδώ, ο οποίος όμως θα μας λέει περισσότερο ε, το τι περίπου θα συμβεί. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ περισσότερο είναι η νομοθετική στρατηγική που θα ακολουθήσουμε γιατί γνωρίζουμε πως ευθύ εξ αρχής είναι ε, πολύ πιο εύκολο πάντα να ε, ξεκινάμε από χαμηλά, αν θέλετε, από ένα χαμηλό επίπεδο ε, εναρμόνισης και μετά είναι δυσκολότερο βέβαια στο μέλλον να κινηθούμε διαφορετικά, δηλαδή να το ανυψώσουμε και πάλι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο στόχο μα. Να δημιουργήσουμε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή σε ό,τι αφορά το επίπεδο προστασία και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να σηκώσουμε, να ανυψώσουμε αυτό το επίπεδο παρότι θα είναι δύσκολο. Μετά είπατε ε, πως ε, σε ό,τι αφορά τη μέθοδο, την ενιαία μέθοδο που θέλετε να ισχύσει, ότι δεν θέλετε να δημιουργήσουμε ένα ε, τέτοιο φραγκενστάιν δηλαδή ένα συνοθήλευμα από διαφορετικά στοιχεία προστασίας, πολιτικών προστασίας. Όμως αυτός ο φραγκενστάιν έχει ήδη δημιουργηθεί. Όταν έχουμε δηλαδή home visit travel events για παράδειγμα, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αυτό αυτό το συνοθήλευμα, αυτό ο Φραγκενστάιν και εκεί πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόμαστε εναρμόνιση αν θα πρέπει να παραμείνει η διαφοροποίηση όσο έχει. Και σωστό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να συγχαρώ την Επίτροπο Κούνεβα για όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει στο παρελθόν και της εύχομαι βέβαια ό,τι καλύτερο ε, και για το μέλλον γιατί οι δράσεις τις οποίες οργάνωσε εκείνη ήταν ε, μερικές από εκείνες που έγιναν δεκτές με το πιο θετικό τρόπο από τους καταναλωτές. Ε, η έκθεση από τις χρηματοδοτικέ υπηρεσίε για του καταναλωτέ που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στου καταναλωτέ τη δική μου χώρα στη Ρουμανία. Ε, βλέπουμε δηλαδή συχνά πως ε, σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή να παρατηρείται ε, ελλειπής διαφάνεια, υψηλό κόστος και ούτω καθεξής. Ζητήματα δηλαδή με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε. Το δικό μου ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πέρα από τις συγκεκριμένε δράσεις που μας αναφέρατε, έχετε οραματιστεί και δράσεις κατά των προβλημάτων όπως αυτά παρουσιάζονται σε σχέση με τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες και επίσης ε, σε ό,τι αφορά τον τομέα των ιατρικών σφαλμάτων και την κακή πρακτική, ε, προβλέπετε να κάνετε κάτι. Γιατί θεωρούμε πως αυτό το ζήτημα δεν είναι αμυγό ζήτημα υγείας, είναι περισσότερο ζήτημα προστασίας και πάλι του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο για την παρουσίασή της και να αναφερθώ σε αυτό που είπε την βελτίωση της εσωτερικής αγοράς. Συγκεκριμένα σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες έχει ζητηθεί μελέτη επιπτώσεων από τα κράτη-μέλη στην οποία όμως δεν περιλαμβάνονται κοινωνικές παράμετροι. Εμείς διαφωνούμε με αυτή τη λογική γιατί υπάρχει σαφής επηρεασμό του εργατικού δικαίου. Κατά την άποψή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στην ανάλυση των επιπτώσεων για την εφαρμογή της οδηγίας να λάβει υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες της οδηγίας σε διαβούλευση πάντοτε με τους κοινωνικούς εντέρους. Τι μέτρα προτίθεστε, κυρία Επίτροπε, να λάβετε. Συνάδελφοι, ευχαριστώ. Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις για σας, κυρία Κούνεβα. Κύριε Κορέια Κάμπος, ο συγκριτικός πίνακας είναι χρήσιμος γιατί διευκρινίζει την κατάσταση για τα δικαιώματα των καταναλωτών δυνάμει της οδηγίας για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Θα αναθεωρήσουμε, θα εξορθολογήσουμε τις τέσσερις υφιστάμενες οδηγίες όπως είχε ζητήσει το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι πολύ ευκολότερα θα πολλούν διασυνοριακά επιχειρήσεις και το ρυθμιστικό περιβάλλον θα γίνει πολύ πιο προβλέψιμο και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις επίσης Επίσης, μία, ε, με ρωτήσατε για την πολιτική. Όχι, δεν σας ζητώ να το πίστευε και μία ερεύνα. Υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία και θα συνεχίσω να σας τα δίνω. Το μόνο που σας ζητώ είναι να έχετε ανοιχτό πνεύμα και να βλέπετε ε, τη σφαιρικότερη εικόνα. Τι θα γίνει με την ε, ψηφιακή αγορά της οθόνης αν είναι κατακαιρματισμένη. Τι θα γίνει αν δεν έχουμε αυτή την οδηγία που προσανατολίζεται προς την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις. Ξέρετε τι εννοώ. Είναι το γιν και το γιάνγκ της ίδιας αγοράς. Ε, γι' αυτό στην κρίση μας είναι τώρα. Πώς ε, θα οικοδομήσουμε μια αγορά άνετη και συμπληρώνει τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η αγορά. Υπάρχει επιχειρηματική πλευρά της οδηγίας, ε, αλλά ανέκαθεν ναι, είχα και την άλλη πτύχη ε, στο μυαλό μου. Γιατί αν υπάρχει συμφόρηση στις, αγο... στις αγορές ε, λόγω των υπεράριθμων κανόνων η... το αποτέλεσμα δεν θα είναι θετικό για τους καταναλωτές. Θα συνεχίσουμε το διάλογό μας και θα σας ενημερώνω ε, διαρκώς και θα διαβουλεύομαι μαζί σας για να με πιστέψετε, για να πιστέψετε ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα για το μέλλον. Ε, κύριε Σορ, για τις ιατρικές υπηρεσίες, το scoreboard, ο πίνακας βαθμολογίας για τους καταναλωτές μας βοηθάει για να ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας και κάνουμε και άλλες αναλύσεις, στις μεταφορές, στην ενέργεια στις τράπεζες. Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι πιο εξειδικευμένες. Η αρμόδια επίτροπος ε, εργάζεται με εξαιρετικό τρόπο ε, και έχει, έχει τοποθετηθεί Αλλά καλά κάνετε και κρούετε τον κόδωνα του κινδύνου. Θα δούμε από πού προέρχονται οι περισσότερες καταγγελίες. Να άλλο ένα από τα ωφέλη της ε, οδηγίας. Ε, ονειρεύομαι την ημέρα όπου ε, θα χρησιμοποιούμε τις καταγγελίες για να νομοθετούμε, ε, δηλαδή να ξέρουμε τι θέλουν οι άνθρωποι. Εκείνοι σφιγμομετρούν την αγορά και χάρη σε αυτούς μπορεί να λειτουργήσει αισίως η αγορά. Το τελευταία ερώτηση για την CRD. Ε, έκανα ε, εκ βάθους μελέτη αντίκτυπου και συμπεριέλαβα και τον κοινωνικό αντίκτυπο της οδηγίας ε, ε είναι θετικά τα αποτελέσματα γιατί ε, χάρη στην οδηγία θα απελευθερωθεί η εσωτερική αγορά και θα υποφεληθούν οι καταναλωτές, θα έχουμε καλύτερες τιμές και καλύτερης ποιότητας ε, υπηρεσίες και προϊόντα επ' αυτού θα βασίσουμε την εσωτερική αγορά να ε, εστιάζεται γύρω από τον καταναλωτή. Ε, φτιάξαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Τώρα ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε τις ανάγκες των πολιτών, των καταναλωτών. Αυτό είναι το νέο βήμα. Με συμμετοχική οικονομία θα αλλάξει η κατάσταση. Ε, αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση, κύριε Χάρμπουρ. Έτσι δεν είναι να αποχαιρετήσω τώρα τα μέλη της Επιτροπής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εμπνεύσατε με τα σχόλια για τις παρεμβάσεις σας. Οι ερωτήσεις σας ήταν ορθές, ε, ελπίζω να ήταν και οι απαντήσεις μου και ελπίζω μελλοντικά να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε και πάλι σας ξαναλέω ότι οποτεδήποτε με χρειαστείτε για αυτή την οδηγία, εγώ στη διάθεσή σας είμαι. Ευχαριστώ. Uh, well, I think, um, Επίτροπε, ε, αυθόρμητα σας χειροκροτεί ε, το ακροατήριο. Αυτό δείχνει πόσο χαιρόμαστε όταν έρχεστε και καταδεικνύεται πόσο μεγάλη δέσμευση έχετε αναλάβει και πόσο αφοσιωμένοι είστε. Ακούσαμε 16 συναδέλφους ε, που έθεσαν διεξοδικά ερωτήματα. Ε, η αυτή η οδηγία είναι ύψιστη προτεραιότητα για μας σήμερα και αύριο σας παρακαλώ λίγη ησυχία, λέει ο Πρόεδρος, ε, δείξτε λίγο σεβασμό για την Επίτροπο. Αύριο στις 3 μέχρι τις 6.30 θα κάνουμε διεξοδική συζήτηση για την οδηγία προστασίας των καταναλωτών και όσοι μπλέκεστε στο θέμα αυτό σίγουρα θα είστε αύριο εδώ υπό την ηγεσία του Αντρέα Σουβάπη για να συζητήσουμε και συμφωνήσαμε να εκπονήσουμε ε, γνωμοδότηση σε πρωτοβουλία για το πίνακα βαθμολογίας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με εσά και το επιτελείο σας. Σας Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε μέχρι το πέρας της ε, θητείας σας ε, και ίσως και αργότερα, ποιος ξέρει. Κυρία Ράπτη, διαδικαστικό έχετε? Μία πρόταση. Ε, χαίρομαι πραγματικά και αισθάνομαι την ανάγκη να πω το εξής. Ε, από την Επίτροπο ακούσαμε εκτός από το ρήμα νομίζω, εκτός από το ρήμα θεωρώ και το ρήμα ονειρεύομαι όταν μία επίτροπος χρησιμοποιεί και το ρήμα «ονειρεύομαι», νομίζω ότι ακόμα εμείς ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Thank Σας ευχαριστούμε. Ε, ίσως ε, θα, στην Επιτροπή θα έχουμε και άλλους οραματιστές. Ε, θα έρθετε στις ε, ακροάσεις των νέων επιτροπών. Κυρία Ράπτη, μπορείτε να πάτε στην ακρόαση της, ε, του επόμενου επιτρόπου για τα θέματα των καταναλωτών για να τους ρωτήσετε ποια είναι τα όνειρά τους αυτά για τις επόμενες ανακρίσεις που θα γίνουν. Την επόμενη ιερά εξέταση των επιτρόπων. Ένα ε, διαλυματάκι θα κάνουμε μέχρι να αποχωρήσει η Επίτροπος και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Uh, so, ladies and gentlemen, can we, um, can we resume, please? Uh, if you could take... Συνεχίσουμε, συνάδελφοι, να μπορείτε να καθίσετε στις θέσεις σας για να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Πρωτού, λοιπόν, συνεχίσουμε στο το πολύ σημαντικό σημείο των πεθαμένων πληρωμών payments θα ήθελα να πω δύο λόγια εδώ γιατί δεν έκανα κάποιε ανακοινώσει εδώ καθώ ε, αρχίσαμε κατευθείαν με την κυρία Κούνεβα αφού είχαμε αργήσει. Θα ήθελα λοιπόν ε, καταρχήν να ευχαριστήσω όλου όσου είχαν συμμετάσχει σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αποστολή στη Σουηδία την περασμένη εβδομάδα, στο τη Επιτροπές μα, ο κύριο Σφάμπο, ο κύριο Άρια, κυρία Χέτ, ο κύριο Ταραμπέλα, η κυρία Σαρδεμόζα Κύριε Λούκεγκαρτ, ήταν όλοι παρόντες και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα απελαγή απόψεων σε ό,τι αφορά το τα γενικότερα ζητήματα της προστασίας ε, ε, του καταναλωτή, των δημοσίων προεκτηριών και ούτω καθεξής. Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα από την πλευρά τη στους του δύο συναδέλφου για την πολύ καλή οργάνωση αυτή τη αποστολή, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και το λέω αυτό ε, για τους ε, νέου συναδέλφου εδώ, οι οποίοι ενδεχομένω να ενδιαφέρονταν ε, για να εκδηλώσουν το να, να, να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους αποστολές. Είχαμε δηλαδή πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Σαμπούνη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα προστασία του καταναλωτή. Είχαμε συνάντηση και με τι αρμόδιε αρχέ για την προστασία του καταναλωτή και και τι ε, αρχέ ε, που είναι αρμόδιε για τις ε, δημόσιες προμήθειε Λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύτιμα για τις εργασίε μας. Δεύτερη ανακοίνωση τώρα που θα ήθελα να κάνω. Είχαμε δύο συνεδριάσεις πρόσφατες των συντονιστών. Καταρχήν, λοιπόν, συμφωνήσαμε πως τα σημειώματα των αποφάσεων που θα λαμβάνονται στι συνεδριάσεις των συντονιστών θα διαβιβάζονται σε, όλους, ε, σε όλα τα μέλη τη επιτροπή, ώστε όλοι σας να έχετε δυνατότητα να εξετάσετε σε λεπτομέρεια αυτέ τι αποφάσει, οπότε δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειες απλά ε, ε, εξετάσαμε σε αυτές τις τελευταίες συνεδριάσεις το πρόγραμμα εργασιών μα. Έχουμε ε, συμφωνήσει για τα κυριότερα σημεία ποιοι θα είναι οι εισηγητές ε, και την εκκίνηση εργασιών ε, συγκεκριμένα απάντηση σε τρία ανακοινώσεις των επιτροπών, το Market Scoreboard, το Consumer Scoreboard και την έκθεση Solve. Και επίσης συμφωνήσαμε και επί μια σειρά άλλων εκθέσεων εμπόδια, για παράδειγμα, στην ενιαία αγορά ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αφού παίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο τη ενιαία αγορά, να εξετάσουμε τι νέε εξελίξει στον χώρο των δημοσίων ε, προμηθειών. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν, ε, θα ξεκινήσουν, αρχίσει η κατάρτιση των εκθέσεων και είπαμε να έχουμε αποστολές στην Ισπανία που θα έχει αναλάβει την Προεδρία στην Ινδία για ζητήματα ασφάλεια και, ε, και άλλα θέματα προστασία του καταναλωτή που σχετίζονται και με ζητήματα βέβαια που αφορούν και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Κόρο και άρα σχετίζονται και με τη δική μα έκθεση. Και θα έχουμε ερωτήσει από τη δική μα πλευρά προ το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά ε, την οδηγία για τις, ε, την, για τις υπηρεσίες και ελπίζουμε πως αυτό θα συμφωνηθεί από την πλευρά των Προέδρων ε, πριν από την ημερομηνία ε, που ξεκινάει ή που αρχίζει να τρέχει πλέον θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο που είναι νομίζω 21 Δεκεμβρίου. Ε, μετά ένα, μια επερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το πού βρισκόμαστε, σε ό,τι αφορά τον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και την ερχόμενη εβδομάδα τον Οκτώβριο θα σας παρουσιάσουμε και μια μελέτη σε ό,τι αφορά την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο αυτής της οδηγίας σε ό,τι αφορά δηλαδή τα επαγγελματικά προσόντα γιατί αναφέρθηκαν πολλά προβλήματα εκεί και πιστεύω πως οι συντονιστέ θέλουν να συνεχίσουν να παρακολουθούν αυτό το τομέα. Ένα ακόμα σημείο το οποίο βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη είναι το εξή η κυρία Βιόλινγκ θα ήθελε πολύ να μας ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα το οποίο θα λάβει η χώρα αρχές Δεκεμβρίου. Και επειδή δεν θα μπορέσει να περιβρεθεί σε μια συνέντευξη της Επιτροπής μας, θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε μια τηλεδιάσκεψη, video conference, κατά την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν εδώ να το προβλέψουμε αυτό σωστά με το σωστό χρονοδιάγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές για, την, για το πολύ μεγάλο ενδιαφέροντους ε, για το νέο πρόγραμμα εργασιών μα ε, και να ευχαριστήσω και του αντιπροέδρου εδώ. Ε, θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα λοιπόν και θα έχουμε και τη λήψη επίσημα των σχετικών αποφάσεων και βέβαια με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν και στο πλαίσιο των επόμενων συνεδριάσεων θα υπάρχει χώρος για να συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, τα μέλη δηλαδή της Επιτροπής. Ας περάσουμε τώρα στην δεύτερη ανταλλαγή απόψεων μα γιατί είχαμε καταρχήν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο. Να περάσουμε λοιπόν στην δεύτερη ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά ε, την ε, νέα, αναθεωρημένη δηλαδή, πρόταση τη της ε, Επιτροπή για τι καθυστερημένε πληρωμέ, late payments. Είχαμε, έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μα την κυρία Βάλα, η οποία είναι πολύ πεπειραμένη και σε προηγούμενε επιτροπέ του Κοινοβουλίου ε, ή και αναλάβει και ω εισηγήτρια. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους κοιόδους εισηγητές, η κυρία Χάνσλεκ από το ΑΕΛ και η κυρία Χόντσμαν από την ΑΛΤΕ. Αναμένουμε από τους πράσινους τον διαβισμό ενός ε, εισηγητή, η κυρία Ρούλα. Ο κύριος Κόζεσνικ για το ECR και η κυρία από την ΚΟΕ. Ε, με χαρά μου λοιπόν πιστεύω ότι όλοι οι όλες είναι εδώ. Και βέβαια στη συνέχεια μετά από τις παρεμβάσεις ε, της εισηγήτριας και όλων των εισηγητών, εισηγητών ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε το λόγο και σε όλους που θέλουν να μιλήσουν. Ήθελα να ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος εδώ από την Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων Μηχανίας για να μας ε, για να τοποθετηθεί όχι αλλά έχουμε ε, και τη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα έχει παρουσιάσει τη μελέτη αντικτύπου σε προηγούμενη συνεδρίαση για το ίδιο ζήτημα. Οπότε σα καλωσορίζουμε και πάλι για να σχολιάσετε τα όσα θα ακούσετε από την πλευρά τη Επιτροπή μα. Ο λόγο λοιπόν στην εισηγητή. vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich bin zwar erst seit, äh, Stunden Ορίστηκα λοιπόν ε, πριν από όρους ουσιαστικά ως ε, συγκήτρια, αλλά ήδη έχω λάβει ε, πάρα πολλές επιστολές από ενδιαφερόμενους ε, φορείς, οι οποίοι βέβαια έχουν και πάρα πολύ διαφορετικές απόψεις. Όμως θα επανέλθω σε αυτό. Να πω λοιπόν ότι έχουμε προβεί σε πάρα πολλές ανταλλαγές απόψεων σε ό,τι αφορά τις καταστρέψεις πληρωμών και είχαν τεθεί μια σειρά από θέματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία έχουν παραμείνει αναπάντητα και θα πρέπει να ασχοληθούμε και πάλι με αυτά, αλλά ε, έχουμε ε, εξ αρχής εκδηλώσει την θετική μας στάση ότι δηλαδή θεωρούμε την εν λόγω πρόταση ως ένα ακόμα ε, βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης του γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας και ε, βήμα προς την καταπολέμηση εμποδίων που υπάρχουν ακόμα ε, σε αυτόν τον τομέα που και επιβαρύνουν ιδιαίτερα βέβαια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω και της οικονομικής ε, κρίσης. Και βέβαια, δηλαδή πιο συγκεκριμένα ότι θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες βέβαια θα πρέπει να η ε, ιδιαίτερα ή είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ζητήματα cash flow. Άρα λοιπόν, ε, το ζήτημα των, των καθυστερούμενων πληρωμών είναι ένας, ένα από τα ζητήματα τα οποία πολλές φορές οδηγούν τελικά σε χρεοκοπία της επιχειρήσης. Κατά την πρώτη λοιπόν ήδη συζήτηση είχαμε καταστήσει σαφές ότι τουλάχιστον η δική μου πολιτική ομάδα δεν αντιλαμβάνεται πλήρω γιατί οι εν λόγω κυρώσει θα πρέπει να προβλέπονται μόνο για το δημόσιο και όχι για τον ιδιωτικό τομέα. Η αιτιολόγηση ότι δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα κάτι τέτοιο αποτελεί παρέμβαση στο ε, ενοχικό δίκαιο είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο και αναμένουμε βέβαια με ενδιαφέρον την τοποθέτηση τη νομική υπηρεσία. Ε, δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τομεί. Όπω ανάφερε μόλι τώρα και η Επίτροπο, όπου πράγματι παρεμβαίνουμε και μάλιστα με πολύ δραστικό τρόπο στην εθνική νομοθεσία, στο ενοχικό δίκαιο, Άρα μπορεί να είναι θεμητή μια ρύθμιση εδώ στον κρατικό τομέα, στον δημόσιο τομέα, αλλά προφανώ και η πλειοψηφία των εν λόγω συναρχών πληρωμών αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια νέα συζήτηση εδώ με του αρμόδιου εμπειρογνώμονε. Ε, περνάω τώρα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ήθελα να σα ε, προτείνω. Και εκείνο που θα ήθελα να προτείνω να έχουμε όχι μια επόμενη συζήτηση αλλά μια ακρόαση. Ίσως στις 4 Νοεμβρίου αυτό μου προτάθηκε, όχι μεγάλη εκτεταμένη ακρόαση, μια μήνυα ακρόαση, για να έχουμε και όλοι αρκετό χρόνο μέσα στον Οκτώβριο να ακούσουμε την άποψη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των κλάδων και ε, βέβαια θα ήθελα να ε, συμπεριλάβω εδώ και το λέω θέση εξ αρχή και του κοιόδη εισηγητέ για να μην αρχίσουν λοιπόν εδώ να, να περγάζονται μαζί με κάποιε ενώσει οτιδήποτε. Δηλαδή μαζί να πάμε και να ακούσουμε και να συζητήσουμε με τι ενώσει. Και θα ήθελα να προτείνω πως το πρώτο σχέδιο, η πρώτη πρόταση από τη μας πλευρά να συνταχθεί, να καταρτιστεί μετά από την μήνυα ακρόαση γιατί λέμε ότι μέσα στο πρώτο αυτό σχέδιο έκθεσης θα πρέπει να περιληφθούν και κάποιες, ε, κάποια αιτήματα τα οποία θα πρέπει να έχουν συνδιαμορφωθεί και μέσα από την ακρόαση. Οπότε λοιπόν προτείνω κατάρτιση του, της, ε, του σχεδίου της έκθεσης μετά από την μήνυα ακρόαση και στη συνέχεια βέβαια να συζητηθεί τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου και να εγκριθεί εκείνη την περίοδο από την Επιτροπή μας. Δεν ε, βρισκόμαστε υπό μεγάλες χρονικές πιέσεις, αλλά ήθελα παρόλα αυτά να προχωρήσουμε γοργά και αυτό γιατί, και είναι ένας λόγος αυτός που δεν αναφέρεται συχνά, η, η κλάδη, η ίδια οικονομία το ζήτησε ότι θα ήθελε να υπάρξει κάτι εδώ. Ε, πράγμα το οποίο δεν ε, το αναφέρουν συχνά άλλοι συνάδελφοι που έχουν διαφορετική άποψη. Δηλαδή στο πλαίσιο του Small Business Act είχε αναφερθεί αυτό, ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Δεν υπήρξε δηλαδή μία αντίδραση ε, ότι γιατί αναμειγνύεται και πάλι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, ήταν ένα από τα συμπεράσματα αν θέλετε που ε, από το Small Business Act. Αυτά σε ό,τι αφορά το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα, να πάμε δηλαδή ε, αρχές και τέλη ε, Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια, ανάλογα βέβαια με το πώς θα διαμορφωθεί και η συζήτηση εδώ στην δική μας Επιτροπή. Ε, εγώ είχα θεωρήσει αρχικά ότι γρήγορα θα φτάσουμε σε συμφωνία και θα υπάρξει τελικά μια συνένεση μεταξύ μας, αλλά όπως είπα και ευθύς εξ αρχής τελικά υπάρχει... υπάρχουν αρκετά αμφιλεγόμενες απόψεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί υπέρ και υπάρχουν ε, ε, και κάποιοι οποίοι είναι όμως κατηγορηματικά κατά και γι' αυτό θα ήθελα να τους προσκαλέσω όλους αυτούς σε μια ακρόαση ώστε να ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις. Επίσης θα ήθελα να μου απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα το μπορούσαμε να το κάνουμε και με βάση τα όσα είχαμε συζητήσει κατά την πρώτη συζήτηση με τους εστιώδεις. Ε, δηλαδή ερωτήματα εκεί μας είχαν διαφύγει τα οποία δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να εξετάσουμε και να διαπιστώσουμε. Για παράδειγμα το κατά πόσο έλαβε υπόψη της η Επιτροπή την πρόσφατη απόφαση του 10 ή το γιατί αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προβλέψει κάποιο είδους κυρώσεις για τον ιδιωτικό τομέα. Θα τα ρωτήσουμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσουμε τώρα και βέβαια με χαρά μου αναμένω την συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάλα. Λέω πρόεδρος η ιδέα σα ε, για την οργάνωση μια μήνυ ακρόασης και η κατάρτιση του σχεδίου έκθεση από την πλευρά σα μετά από αυτή την ακρόαση αποτελεί μια καλή ιδέα. Και θα ήμασταν σε θέση να σα διευκολύνουμε να το πράξουμε αυτό. Να δούμε βέβαια και τι θα πούνε και οι ιστιώδει. Η κυρία και έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας πω ότι στο δικό μου κράτος μέλος στα πλαίσια της ε, υλοποίησης ενός ε, Small Business Act συναντήθηκα με εκπροσώπους ε, του κλάδου και είδα ότι είναι κάτι το οποίο, είναι ένα έγγραφο το οποίο το περίμεναν όλοι με ιδιαίτερη ε, ανυπομονησία και χαίρομαι που το συζητάμε σήμερα. Επιτρέψτε μου όμως να ασχοληθώ με ορισμένες πτυχές και ίσως να ζητήσω από την Επιτροπή να μας απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη οδηγία. Ε, έχω την εντύπωση ότι το βασικό πρόβλημα όπως αναφέρεται και στην ανάλυση, στην αξιολόγηση αντικτύπου, έχει να κάνει με με το φόβο που υπάρχει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το ότι θα χάνουν ένα πελάτη, ε, θα χάσουν τον πελάτη. Και βέβαια δεν μπορούμε να του αλλάξουμε νοοτροπία, γιατί δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις αποφάσεις τους. Αλλά κατά την άποψή μου, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που θα τους ε, ε, οθήσουν στο να καταλάβουν τα δικαιώματά τους. Πολύ συχνά, μια μικρομεσαία επιχειρήση, επιχειρήση δεν θα ζητήσει αυτά τα επιτόκια. Γιατί ε, μερικές φορές ε, ε μπορεί να υπερβαίνουν και το φιλόμενο ποσό. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα στη χώρα μου όπου το κόστος μπορεί να είναι υψηλότερο ε, από τα επιτόκια. Το διοικητικό κόστος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όταν μιλάμε για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές. Δυστυχώς, είναι αδύνατο σε πολλές περιπτώσεις σε, αυτό το συγκεκριμένο θέμα ε, να υπάρξει αποζημίωση. Αυτή η νέα νομοθεσία λοιπόν θα αποτελέσει ένα σημαντικό νομικό όπλο στα χέρια των μικρομεσαίων. Αλλά νομίζω ότι περισσότεροι από τους μικρομεσαίους επιχειρήσεις από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη τη νέα νομοθεσία. Πολύ συχνά οργανώσει επιχειρηματιών θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την ε, κατεύθυνση. Γιατί οι οργανώσει των ε, επιχειρηματιών θα μπορούσαν να διαδώσουν αυτέ τι πληροφορίε. Ρωτώ λοιπόν, δεν βλέπετε μια ε, πιθανότητα να υποστηρίξουμε τέτοιε δράσει συνειδητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για, για, να μάθουν για αυτή την υπόθεση των επιτοκίων, για παράδειγμα. Κάτι άλλο το οποίο είναι σοβαρό και θα πρέπει να το δούμε είναι το θέμα της εναρμόνισης των όρων πληρωμής. Νομίζω ότι αυτή, αυτό το χρονικό διάστημα 30 ημερών είναι καλό σημείο εκκίνησης. Από την άλλη βεβαίως καταλαβαίνω ότι Μπορεί οι επιχειρήσεις να δεχτούν, αλλά τα κράτη-μέλη να έχουν αντίθετη άποψη για το θέμα αυτό. Και το πρόβλημά μας ποιο είναι. Ότι αυτό το 5% ως εφάπαξε ως καταποκοπή αποζημίωση. Αυτός ο κανόνας λοιπόν μπορεί να πρέπει να το ξαναδούμε. Πρέπει να απαντήσει η Επιτροπή γιατί υπάρχει αυτό το 5%. Δηλαδή δεν αμφισβητώ το μέσον, αλλά γιατί 5%. Ίσως λοιπόν εδώ θα μπορούσε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διαφωτίσει. Και κάτι άλλο αναρμόνιση πληρωμών όταν πρόκειται για συναλλαγή ανάμεσα σε επιχειρηματίες. Όταν η προθεσμία πληρωμή συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση, γιατί εδώ πρέπει να το δούμε το θέμα και να μην παρεμβαίνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον ε, υπάρχει αυτή σαφώς η επιθυμία, από όλους δηλαδή η επιθυμία για εναρμόνιση της προθεσμίας. Και κάτι άλλο. το ειδικό καθεστώ για τι πολύ μικρέ επιχειρήσει όσον αφορά τι καθυστερημένε πληρωμέ. Δυστυχώ στην αξιολόγηση αντικτύπου δεν αναφέρεται τίποτα για το θέμα αυτό. Και από ό,τι θυμάμαι, οι περισσότεροι από τι συμμετέχοντε στη διαβούλευση τάχθησαν υπέρ τέτοιου είδου λύσεων. Θέλω λοιπόν η Επιτροπή να μα δώσει ορισμένε πληροφορίε και βεβαίω ελπίζω να συνεργαστούμε ιδιαίτερα προοικοδομητικά με τον εισηγητή και χαίρομαι ιδιαίτερα και ε, με τη δημόσια ακρόαση και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ακούσουμε την άποψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από την Πολωνία. Σε ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για την ε, ε, συνολική σας τοποθέτηση για το θέμα. Ξέρω ότι είστε και ίδια επιχειρηματίες, έχετε μια μικρομεσαία επιχείρηση και καταλαβαίνω ότι σας καίει το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών. Ε, αργότερα θα τοποθετηθεί και η Επιτροπή σε όλα αυτά τα ζητήματα ε, τα οποία ανέφερε και ο συγητή και οι σκιώδει συγητέ. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κότσμαν που είναι νέο μέλο τη Επιτροπή, δεν έχει ακόμα πάρει το λόγο. Ε, Σα παρακαλώ να τοποθετείτε εκ μέρου εμά του φιλελευθέρων. Ο κύριο Κρότσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί της αρχής ε, ε, χαιρετίζουμε μια τέτοια πρόταση οδηγία, ε, γιατί δίνει ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους τύπο μονοπωλίων, για παράδειγμα δημόσιες επιχειρήσεις, κοινότητες και ούτω καθεξής. Αλλά από την άλλη πλευρά ε, γνωρίζω, γιατί και εγώ ήμουνα για πολλά χρόνια ενεργό στο τομέα ακριβώ τη ε, τοπική αυτοδιοίκηση, οι δημόσιε αρχέ οι οποίε ε, προβαίνουν πολύ έγκαιρα στι δικέ του πληρωμέ. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις κάθε φορά. Υπάρχουν δηλαδή δημόσιες οι υπηρεσίε των οποίων οι υπάλληλοι αφήνουν απλά κατά μέρο κάποια τιμολόγια και τα εξοφλούν απλώ αργότερα. Ε, τέθηκε το ερώτημα το γιατί γίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ ιδιωτικών ε, και δημοσίων ε, φορέων εδώ. Στι δημόσιε αρχέ έχουμε για παράδειγμα δήμου και κοινότητε που έχουν συγκεκριμένο ταμείο και μπορούν ανα πάσα στιγμή να προβούν σε πληρωμή. Ε, γιατί μπορούν να λάβουν αυτά τα χρήματα κάθε φορά από τις τράπεζες. Όμως, αν κάτι τέτοιο ισχύσει για, το ιδιωτικό τομέα, ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υπάρξουν προβλήματα, ειδικότερα αφού το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι συχνά μικρό. Ειδικότερα λοιπόν, εάν προβλέψουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή 30 ε, ημέρες ως προθεσμία και μετά 5% ε, είναι πολύ ε, υψηλό το ποσό. Δηλαδή, αν προβούμε σε συσσωρευτικό υπολογισμό, μιλάμε για 60%, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ε, υψηλό βέβαια αυτό το ποσό και θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο είναι ε, θεμητό ή είναι σκόπιμο εν να επεκτείνουμε τέτοιου είδους διατάξεις σε όλες ανεξαρτήτως τις ιδιωτικέ επιχειρήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλουμε να, να έχουμε και εδώ τρόπους διασφάλισης της έγκυρης πληρωμή. Ε, συχνά έχουμε στο πλαίσιο ε, συμφωνιών συγκεκριμένους όρους επιπληρωμής οι οποίοι προβλέπονται και νομίζω πως ε, οι, τα, οι όροι αυτοί που προβλέπονται στο πλαίσιο του, το ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ισχύουν και αντίστοιχε υποχρεώσει. Θα ήταν καλό να ισχύουν αντίστοιχε υποχρεώσεις με αυτές στο δημόσιο τομέα. σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος για την εισπράξη, ε, δεν ξέρω γιατί εδώ έχουμε διαφοροποίηση. Δηλαδή το κόστος είναι ίδιο, είτε έχουμε να κάνουμε ποσό χιλιών ευρώ είτε με 100.000 ευρώ. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί πρέπει να έχουμε διαφορετικά ποσοστά και να θέτουμε αυτό το όριο πάνω από τα 10.000 ευρώ ή όχι. Ε, δεν γνωρίζω δηλαδή κατά πόσο έχει νόημα να υπάρχει μια τέτοια διαβάθμιση. Ε, κυρία Βάιλα, εμεί είχαμε μια σύντομη συζήτηση. Εντάξει, όταν λέω εμεί εννοώ εσεί με εμά την άλλη αλλά για, εκείνους, ε, για εκείνες επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε εξαγωγές σε άλλα κράτη-μέλη ε, θα είναι μια τέτοια διάταξη πολύ ωφέλιμη γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βέβαια εξάγουν σε χώρες με διαφορετικούς όρους πληρωμής και μια τέτοια οδηγία ακριβώς θα προωθούσε την ενιαία άκορα. και προφανώς και τη χαιρετίζουμε με αυτή τη συλλογιστική. Υπάρχει βέβαια και μια ακόμα συζήτηση εδώ, δηλαδή το κατά πόσο η ε, κυρώσεις αυτές για τις ε, καθυστερήσεις ε, πληρωμών συνιστούν κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι το άγνωστο στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, αλλά αποτελεί ένα τρόπο ή ένα επιχείρημα προκειμένου και οι δημόσιες αρχές να τηρούν ακριβώς αυτήν την προθεσμία περί εξόφλησης δηλαδή των 30 ημερών. Ε, το γεγονός ότι έχουμε 30 ε, ημέρες ε, μας δείχνει ότι πράγματι είναι και δυνατή η σχετική εξόφληση από την πλευρά των δημοσίων επιχειρήσεων. Μάλιστα έχουμε το ειδικότερα από την πλευρά των μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων. Ε, μηχανοργάνωση εδώ ε, όπου όλα γίνονται ηλεκτρονικά και αυτόματα και εγώ επειδή σας λέω πως βρισκόμουν σε τέτοιου είδους ε, ε, δημόσιες αρχές είδα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως εκείνο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η ρευστότητα και στις μικρόνες επιχειρήσεις θα πρέπει να το δούμε αυτό. Από τη μία δηλαδή όταν κάποιο αναμένει να εισπράξει κάποια χρήματα, τότε βέβαια θέλει να τα εισπράξει το ταχύτερο δυνατό. Αλλά από την άλλη, όταν είναι ο φιλέτη, διαφοροποιείται η κατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί να μην έχουμε εδώ ακριβώς την ίδια μεταχείριση για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ίσως θα πρέπει να ισχύουν δηλαδή και διατάξεις στο πλαίσιο των ε, συμβάσεων. Ε, ε, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας επειδή ακριβώς πρόκειται για μια νομοθεσία η οποία πρόκειται να ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη. όπου ε, για παράδειγμα έχουμε μεγάλες ε, διαφορές. Δηλαδή, ε, όπως είπε μόλις τώρα και ο συνάδελφος κ. Μπουσά, στη Ρουμανία έχουμε κάποιες δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν και νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Λαμβάνουμε όμω και ταυτόχρονα υπόψη, όπω υπόθηκε και από πλευρά τη Επιτροπή, ότι με, μια ε, τέτοια ρύθμιση θα είχαμε βέβαια μια, ε, σημαντικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την αύξηση τη δευσότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Η κυρία Ρούλε. Ε, πολύ σύντομα να πω πω ε, και εμεί χαιρετίζουμε αυτή την οδηγία, αλλά χαιρετίζω και το γεγονό ε, ή μάλλον τη δήλωση τη κυρία Βάιλερ ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα γιατί πολύ συχνά εδώ το πρόβλημα βρίσκεται στη λεπτομέρεια και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ειδικότερα για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τι 30 ημέρε, Το ζητούμενο είναι ε, να διασφαλίσουμε να, είναι, ε, ε, να έχουν υποβληθεί όλα τα σχετικά έγγραφα. Γιατί για τη δημόσια αρχή είναι πάντα απαραίτητο αυτό να έχει λάβει τα απαραίτητα έγγραφα που προβεί στην πληρωμή. Ή για παράδειγμα αν υπάρχουν κάποια ελαττώματα, ε, στην οποία περίπτωση ο φιλέτης ε, δεν προβαίνει στην πληρωμή μέχρι να υπάρξει μια επίλυση αυτών των ελαττωμάτων ή προβλημάτων. Ε, και επίσης θα πρέπει να γίνει και μια θεμελιώδη συζήτηση σε ό,τι αφορά αυτό το, το, το ποσοστό του 5% γιατί κάτι τέτοιο ουσιαστικά τελικά δεν αποτελεί αποζημίωση, αποτελεί κύρωση, αποτελεί τιμωρία. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να περιλάβουμε τέτοιου είδου τιμωρία εντό εισαγωγικών σε μια τέτοια οδηγία. Εμεί είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά βέβαια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συζητηθεί εκτενώ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που άκουσα ε, την ημερομηνία τον Νοέμβριο γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες ε, πληροφορίες. Συμφωνώ με την ε, κυρία Βάιλερ. Αυτή η πρόταση μας ε, μιλάει για διαφόρων ειδών επιχειρήσεις. Αυτές προμηθεύουν τον κρατικό τομέα και οι υπόλοιπες. θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται ρύθμιση και στον ιδιωτικό τομέα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο προκλητικά, να αναφερθώ στον κανονισμό που ήδη υπάρχει σε αυτό το τομέα. Ε, μπορούμε να επιβάλλουμε την καταβολή των πληρωμών. Υπάρχει σχετική οδηγία που άρχισε να ισχύει πριν από μία πενταετία. Δεν ε, Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ρύθμιση, γιατί αυτό δεν συνιστά έχει για την ε, εύρυθμη λειτουργία των κανόνων. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αξιολόγηση αντικτύπου ε, επί του, των κρατικών κονδυλίων Συνεπάγεται κόστος ε, αυτή η οδηγία και πρέπει οπωσδήποτε να υπολογιστεί αυτό το κόστος. Πέρα από τις κυρώσεις και τις ποινές, νομίζουμε ότι η πρόταση αυτή ανοίγει το παράθυρο για μεγαλύτερη διαφθορά. Σας ευχαριστούμε ε, για τις παρατηρήσεις σας. Ας μας μιλήσει λοιπόν η Επιτροπή και για το κόστος που αυτό συνεπάγεται. Ο κύριος ε, Τζιόν για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικές οι λεπτομέρειες μέσα στην πρόταση αυτή. Έχουμε ακούσει σχόλια από διάφορες ε, οργανώσεις. και σχετικά με την αρχή της ε, συναλλαγής, ε, ε, αν δεν συμπίπτει η ημερομηνία της συναλλαγής με την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, θα έπρεπε να συζητήσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να συζητήσουμε σε επόμενη συνεδριά που λέει η κυρία Βάιλερ. Πάντως, θα ήθελα ήδη σήμερα μια απάντηση από πλευρά τη Επιτροπής για το εξή. Υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα, λαμβάνοντας υπόψη και την επικουρικότητα, ε, ε, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι ε, παρεμποδίζεται ουσιαστικά η ελεύθερη κυκλοφορία. Θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση ανάμεσα στον ε, δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί κανείς να προτάξει το επιχείρημα της επικουρικότητας ε, ακόμη και στις σχέσεις B2B από επιχείρηση προς επιχείρηση. Πάντως ε, βρήκαμε ε, ότι δεν διευκρινίζει την κατάσταση η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλα αυτά θα δείξουμε ανοιχτό πνεύμα. Ευχαριστούμε όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, και σίγουρα θα γίνουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις γιατί υπάρχει πληθώρα απόψεων για το θέμα και καλό είναι αυτό, προάγει το διάλογο. Η κυρία Στήλερ και μετά να κλείσουμε προτείνω τον κατάλογο των ομιλητών γιατί δεν έχουμε πια χρόνο στη διάθεσή μας. Κυρία Στήλερ, Ευχαριστώ. Στάιλερ, Στάιλερ ε, ονομάζομαι, σας διορθώνω την προφορά για μελλοντική χρήση. Έλεγα λοιπόν ότι συγχαίρω την Μπάρμπαρα που ανέλαβε το ρόλο της συγγήτριας. Είναι σωστή η προσέγγιση σου και ε, μου αρέσει ε, ότι προτείνεις διάφορες ακροάσεις. Για τα επιμέρους ζητήματα Α πάρω το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι τοπικές αρχές σε ποσοστό 93% των τιμολογιών εξασφαλίζει πληρωμή μέσα στι 30 ημέρε. και το θέμα του καταποκοπή ποσού και του κόστους ανάκτησης των ποσών φαίνεται απαγορευτικό για κάποιες ε, τοπικές αρχές, αλλά ήδη εργάζονται καλά και έχουν καλά αποτελέσματα για την ημερομηνία πληρωμή. Σε Μπάρμπαρα, αυτό το θέμα του 5% για τις καθυστερημένες πληρωμές, αυτό δεν εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Υπάρχει και το θέμα των τιμολογίων που αποστέλλονται σε λανθασμένη διεύθυνση κτλ. Μπορούμε, χρησιμοποιούνται νέα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πλειοψηφία των καθυστερούμενων πληρωμών προέρχονται από άλλε επιχειρήσεις και όχι από τον κρατικό τομέα. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το ζήτημα των ε, ε, καθυστερημένων πληρωμών έχει μέγιστη σημασία, αλλά χρειαζόμαστε και την ευκαιρία και το χρόνο για να κάνουμε σωστά τη ρύθμιση του τομέα και την έχουμε την ευκαιρία και να αξιοποιήσουμε. Οι τοπικές κρατικές αρχές ε, δεν είναι αυτές προς το παρόν που φαίνουν την ευθύνη για την ημερομηνία πληρωμής ε, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί να τους προσάπτουμε όλα αυτά σε τέτοια ε, περίοδο οικονομικής κρίσης. Σε πάση περιπτώσει καλωσορίζουμε την έκθεσή σας και θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας ερχόμενους μήνες. Σας ευχαριστούμε κυρία Στήλερ, Στάιλερ λέει, ο πρόεδρος Στήλερ. Κάθριν σε φωνάζω βέβαια συνήθω γι' αυτό δεν το θυμόμουν. Στάιλερ, Στάιλερ. Ε, στο μέλλον δεν θα το ξαναπροφέρω λάθος. Η κυρία Μπρίγκμαν εδώ από την Επιτροπή θα θέλατε να σχολιάσετε κάποιες από τις παρεμβάσει. Φυσικά θα έχουμε και πολλαπλές ευκαιρίες στο μέλλον για να το συζητήσουμε το θέμα. Ε, ίσως μετά να ακούσουμε και τη σύνοψη της κυρία Βάιλερ. Αλλά έχουμε ακούσει διάφορε παρεμβάσει. Κυρία Μπρίγκμαν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, που τοποθετήθηκαν. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης ηγητές. Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με την ε, σημασία που αποδίδεται στη λεπτομερή ανάλυση της πρότασης. Ε, πρέπει να αφιερώσουμε τον βετούνο χρόνο για να κάνουμε μια σωστή ανάλυση και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που θα συμμετάσχουμε στη μήνυα ακρόαση που θα προτείνει να οργανώσει η κυρία Βάιλε στις 4 ε, Νοεμβρίου. Ε, είμαστε στη διάθεση της κυρίας Βάιλε και των λοιπόν εισηγητών για να απαντήσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε όλες τις ερωτήσεις σας ε, σήμερα και μελλοντικά στη, στη μήνυα ακρόαση και σε άλλες ε, συνεδριάσεις. Λοιπόν, πολλά από τα σχόλια που ακούσαμε για να απαντηθούν ε, χρειάζεται να επανέλθουμε στη μελέτη αντικτύπου. Εκεί, εκεί βρίσκουμε πολλές απαντήσεις ε, στα ερωτήματά σας. Ακούστηκε η εξής ερώτηση. Είναι σημαντικό να ε, κοινοποιούμε τα πλεονεκτήματα και τα δικαιώματα που προσφέρει στις ΜΜΕ η κοινοτική νομοθεσία για να ε, πληρωθούν ε, οι τόκοι δουλευμένων. Ε, και έχουμε διάφορα μέσα στη διάθεσή μας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων, διάφορα δίκτυα υποστήριξη ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών είναι πολύ σημαντικό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Έχουμε όμω στη διάθεσή μα όλα τα απαιτούμενα μέσα ε, για να ε, ενημερώνουμε με άμεσο τρόπο τις επιχειρήσεις μέσα από αυτά τα δίκτυα και όλοι όσοι χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες ε, μπορούν να τις έχουν χάρη σε αυτά τα μέσα. οποιοδήποτε μέσο υποστήριξης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, δύναται να χρησιμοποιηθεί στο μέτρο που υπάρχει. Έχουμε και την πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί υπάρχουν διάφορες προβλέψεις. Το θέμα ήταν να δούμε αν για τις μικροεπιχειρήσεις ε, μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αυτό το θέμα ε, το εξετάσαμε προσεκτικά και προέκυψε και στη δημόσια διαβούλευση που κάναμε και μέσα στη μελέτη αντικτύπου συγκεκριμένα έχουμε τον πίνακα 223 όπου ε, βλέπετε την άποψη των ε, επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη διαβούλευση ε, σχετικά με το τι χρειάζεται να γίνει. Δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται επιπρόσθετη δράση για τις μικροεπιχειρήσεις. Ε, επιπρόσθετη σχέση με αυτά που ήδη έχουν γίνει γενικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλες ερωτήσεις ε, σχετίζονται με το λόγο για τον οποίο έχουμε διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετική μεταχείριση για τις, επιχειρή... για τις σχέσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις B2B και αφενός και αφετέρου ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα. Είναι σημαντικό να έχουμε την αρχή της συμβατικής ελευθερίας. Είναι μια βασική αρχή του δικαίου και περί συμβάσεων και θέλουμε να τη διασφαλίσουμε αυτή την αρχή και καλό είναι να εναρμονιστούν οι περίοδοι πληρωμής στις ε, συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Αλλά αυτό δεν συνάδει με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα πάντα. Ε, θα κάνουμε μια λεπτομερέστερη παρουσία στη μήνυα ακρόαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ε, πιστεύουμε, να ε, συνειδητοποιήσουμε αυτή τη διάκριση που γίνεται επί τη βάση της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας έχει εξεταστεί η πρόταση από αυτή τη σκοπιά της αναλογικότητας και της επικουρικότητας από διάφορα εθνικά κοινοβούλια. Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Όσα ε, κοινοβούλια έχουν τοποθετηθεί, συμφώνησα με την Επιτροπή ε, ως προς την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας βέβαια ε, μπορούμε να επανέλθουμε και να συζητήσουμε λεπτομερέστερα αυτό το θεμελιώδε ζήτημα. Ε, το θέμα του 5% και της καταποκοπή αποζημίωσης που φαίνεται σαν να είναι μια ποινή ε, σε περίπτωση καθυστέρηση στην πληρωμή που και θα επιβάλλεται από τις δημόσιες αρχές. Λοιπόν, η Επιτροπή κρίνει ότι είναι ε, αρκετά αποτρεπτικό αυτό το ποσό χωρίς να είναι υπερβολικά υψηλό για να μην λοχεύει και αυτός ο κίνδυνος της διαφθοράς που ανέφερε ένας από τους συναδέλφους σας. είναι προσυζήτηση το θέμα σαφώς αν, είναι το σωστό, αν ορίστηκε σωστό επίπεδο αυτό το ποσό, αν ε, γιατί ο στόχος μας είναι να έχουμε τις ε, καλές προϋποθέσεις ώστε να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές ε, οι οι δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό το ζήτημα για ε, το μέλλον. Άλλα ζητήματα τώρα που σχολιάσατε. Η σημασία του να προβλέψουμε μέσα στην οδηγία ε, ορισμένα ποσά για τα, το κόστος ανάκτησης είναι καινοτόμο στοιχείο με βαρύτητα μέσα στην οδηγία. Προβλέπεται μια κλίμακα μέσα στο σχετικό άρθρο. Πάντως, το ότι θα υπεριέχει η πρόταση αυτό το νέο στοιχείο είναι κάτι που καλωσόρισαν οι οικονομικοί φορείς γιατί ε, συνιστά για αυτούς ένα μέσο άμυνα. Στο θέμα της κλίμακας των ποσοστών τώρα, μέσα στην πρόταση του άρθρου 4, ε, θα αποτελέσουν ε, αντικείμενο συζήτησης και φυσικά θέλουμε να γνωρίζουμε και πώς τοποθετήσετε εσείς για αυτό το ζήτημα. Άλλο θέμα, αξιολόγηση του κόστους για το δημόσιο προϋπολογισμό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι διατάξεις. Τα σχετικά στοιχεία τα βλέπετε στη μελέτη αντικτύπου, βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία. Ναι στη μελέτη αντικτύπου έχουμε, έχετε όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Αν τώρα έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις θα πρέπει να κάνουμε πολύ περίπλοκες ε, έρευνες γιατί σε αυτό το τομέα δεν υπάρχουν ε, και ε, αμέτρητα στατιστικά στοιχεία. Αυτά, Πρόεδρε, προς το παρόν και τονίζουμε ότι είμαστε στη διάθεση των εισηγητών ε, και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή τους ε, για να συνεργαστούμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ήσασταν ε, πληρέστατοι τις απαντήσεις και θα θέλαμε να σας ξαναδούμε στο μέλλον σύντομα. Ο κύριος Κάνσπερτ από την Προεδρία είναι εδώ, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας. Δεν θα σας ε, καλέσω να ε, μιλήσετε. Απλά χαιρόμαστε που ε, είσαστε μαζί μας εδώ και παρακολουθείτε τη συζήτηση. Κυρία Βάιλερ, έχετε να κάνετε κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ε, πρόεδρε, ούτως άλλως συνήθως δεν λέω πολλά. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα σχολίασαν και τι απαντήσει που μα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τη μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την ακρόαση, γιατί σίγουρα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσε λεπτομέρειε. Αλλά εκείνο το οποίο δεν βρήκα εγώ μέσα σε αυτή τη μελέτη αντικτύπου είναι τα statements, οι δηλώσει δηλαδή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και προφανώ ω Γερμανίδα κάτι τέτοιο με ενδιαφέρουν πάρα πολύ παρότι ε, δεν υπήρξε μια τέτοια δήλωση από την ε, πλευρά του δικού μου ε, κοινοβουλίου, αλλά σίγουρα η Δανία θα έχει κάνει κάτι, η Αυστρία θα έχει μια δήλωση, οπότε θα θέλαμε να δούμε κάτι. Και να ευστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε κάτι ακόμα εδώ. Όταν λέμε ότι η εμπρόθεσμη καταβολή της πληρωμής ενδεχομένως να είναι δύσκολη για ορισμένες μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να ε, αντιληφθούμε το όλο σύστημα αυτό σε ένα σύστημα το οποίο πρέπει να ισχύει το fair play. Δηλαδή το να μην πληρώνει κάποιο ε, στην ώρα του σημαίνει ότι δημιουργεί προβλήματα σε εκείνον ο οποίο αναμένει αυτή την πληρωμή. Δηλαδή χρειάζεται εδώ ένα fair play και τα προβλήματα ρευστότητα μετακινούνται σε άλλον. Τον προμηθευτή για παράδειγμα ή ε, τον απελάτη. Οπότε το κατά πόσο το 5% είναι υπερβολικά υψηλό ή είναι το κατάλληλο θα πρέπει να συζητηθεί, αλλά κυρώσεις σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν. Οι κανόνες υπάρχουν ήδη. Εάν δεν μπορούμε να ε, ε, καταστήσουμε πιο αυστηρούς τους κανόνες που έχουμε ήδη ή δεν τους κάνουμε πιο ουσιαστικούς, δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε, τότε δεν έχει και νόημα να υπάρχει μια αναθεώρηση της οδηγίας. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε και ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Well, thank Εμείς σας ευχαριστούμε, ιδιαίτερα κυρία Βάιλερ. Να κάνουμε την εξής πρόταση, αν συμφωνείτε. Την επόμενη Τρίτη, όταν θα ξανασυνδριάσουμε, το πρωί και το απόγευμα, μέχρι τότε θα μπορούσατε να μας ε, ε δώσετε μια ένδειξη για το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα χρόνο ακρόαση λοιπά σε διαβούλευση με του κοιόδε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα. Η γραμματεία είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί σα στο θέμα αυτό. Εκτό κι αν ε, έχετε διαφορετική άποψη. Εγώ πάντω νομίζω ότι είχαμε συνολική διάσταση, ε, ε, ανταλλαγή απόψεων. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω. Εκτό και αν θέλετε εσεί για την επόμενη εβδομάδα να βάλετε συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στις, την, την Τρίτη, λοιπόν, στι 6 θα σα δώσουμε ε, ε, χρόνο το πρωί, μόλι αρχίσουμε. Κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ όλου του ηγητέ, του σκιώδει, ε, εκπρόσωπο τη Επιτροπής, ε, του Συμβουλίου. Ως συνήθως, ε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα Ζερμινή και εμείς ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Σας καλούμε αύριο το πρωί στις 9. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Λίγη